Αγαπητοί συνάδελφοι, νομίζω πως δεν σας έδωσα κάποιο χρόνο για να τα πείτε και μετά τις διακοπές, αλλά μπορούμε πια να ξεκινήσουμε. Ελπίζω να περάσατε καλά στις διακοπές σας και ελπίζω να έχετε γυρίσει γεμάτη ενθουσιασμό και ενέργεια για να περάσουν και οι επόμενοι μήνες πριν ξανά κουραστούμε και χρειαζόμαστε και πάλι διακοπές για τα Χριστούγεννα. Λοιπόν, τι μου λένε εδώ οι σημειώσεις μου, πως είναι Τετάρτη 12 Ιουλίου και το ρολόι μου λέει ότι είναι 6 και 19. Ε, πάση περιπτώσει νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε με την ημερήσια διάταξη. Αν δεν υπάρχει καμία τροποποίηση από εσάς, εγώ δεν έχω κάτι, ωραία. Μπορούμε λοιπόν να περάσουμε στις ανακοινώσεις. Αύριο το πρωί θα γίνει μια ακρόαση, μια κοινή ακρόαση για την αναπτυξιακή βοήθεια, που είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα Έχουμε τη σχετική ανακοίνωση Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δυστυχώ, εγώ αύριο το πρωί δεν θα μπορώ να είμαι, γιατί χρειάζομαι να γυρίσω στην ε, περιφέρειά μου, μια και έχω κάποιε υποχρεώσει εκεί. Ελπίζω πάντω πω εσεί θα πάτε. Σα το υπενθυμίζω, θα έχουμε πολλού ε, ομιλητέ και ελπίζω, συνάδελφοι, να έρθετε και να την παρακολουθήσετε. Επίση, την επόμενη εβδομάδα, στι 7 Σεπτεμβρίου, την επόμενη Πέμπτη λοιπόν, η ΣΤΟΑ ε, οργανώνει μία υψηλού επίπεδου ε, συνάντηση ε, για την τεχνολογική καινοτομία, για την ανθρωπιστική βοήθεια και την βοήθεια προς τις πιο ευάλωτες ομάδες. Νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον έτσι ώστε να δούμε πώς μπορούμε μέσω τεχνολογικής πρόοδου, να προσφέρουμε αναπτυξιακή βοήθεια σε όσους το χρειάζονται το ο, συντομότερο δυνατόν. Λοιπόν, αυτή θα γίνει την επόμενη Πέμπτη, 2 με 5.30 και ελπίζω ε, κάποιοι να μπορούν να την παρακολουθήσουν. Άλλες ανακοινώσεις δεν έχω. Μπορούμε να περάσουμε λοιπόν στα πρακτικά της προηγούμενης συναντήσεως 26 Ιουνίου στο φάκελό σας. Αν έχετε παρατηρήσεις προς τη γραμματεία παρακαλώ και αν δεν έχετε θα θεωρήσουμε μέχρι το τέλος της συνεδρίας πως έχουν εγκριθεί. Τέσσερα ανακοινώσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ελπίζω και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πέρασε καλά. Λοιπόν, βλέπω πως έχετε μια ανακοίνωση να μας κάνετε. Ευχαριστώ πολύ. Μια πολύ σύντομη ενημέρωση. Υπάρχει ένα σημείο που ξέρω πως σας είναι ιδιαίτερα προσφυλές. Είναι το σχέδιο δράσης ε, υπαριθμών 2 για το Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο. Χτες ε, ανακοινώθηκε επισήμως είναι η ισότητα των φύλων, η χειραφέτηση των γυναικών και η σχετική ε, στόχη και τα όσα θα συμβούν στην περίοδο 16-20. Επισήμως λοιπόν βρίσκεται και στα δικά σας ε, ε, γραφεία και με μεγάλη χαρά, μια που πλέον ανακοινώθηκε, μπορούμε να το συζητήσουμε και να κάνουμε μια ανταλλαγή απόψεων σε επόμενη συνεδρίαση για όσα ε, σας απασχολούν σχετικά με το θέμα αυτό. Πολύ καλό αυτό και είναι την κατάλληλη στιγμή που παρουσιάζεται. Σήμερα το απόγευμα έχουμε μια ομάδα εργασίας ε, που θα μιλήσουμε με τρεις πρέσβεις και θα σχολιάσουμε το θέμα αυτά. Έχουμε και μία συνάντηση με την Επιτροπή Γυναικών, οπότε με μεγάλη χαρά θα τα συζητήσω όλα αυτά. Βέβαια δύσκολο χρονικά ε, να το τοποθετήσουμε στην ημερήσια διάταξη ή ίσως λοιπόν μα στη μεικτή επιτροπή που θα κάνουμε, συνεδρίες που θα κάνουμε την Επιτροπή Γυναικών να συζητήσουμε και το θέμα αυτό και ε, μάλιστα να το συνδυάσουμε με το χρονοδιάγραμμα για την έκθεση την οποία εγώ ετοιμάζω. Σας ευχαριστώ πολύ. Μπορούμε τώρα να περάσουμε στο σημείο 5 που είναι και αυτό ένα θέμα πολύ σημαντικό για τη δική μας Επιτροπή είναι η εφαρμογή ε, του Trust Fund για την Αφρική, του καταπιστεύματος λοιπόν και να σας πω πως ο πλήρες, ε, ο πλήρης τίτλος είναι ε, αυτό τον οποίο βρίσκεται στα χαρτιά σας και ο οποίος περιγράφει όλους τους στόχους που είναι ακριβώς ε, να καλύψουμε τους ε, στόχους της Βαλέτα το, ε, από τον Νοέμβριο του 2015. Έχουμε ήδη ε, ε, δεσμεύσει 2,8 δις από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης και κάποια βέβαια προέρχονται και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων. Εδώ λοιπόν εμείς έχουμε το δικαίωμα εξέτασης και όταν δημιουργήθηκε το καταπίστευμα αυτό θα θυμόσαστε πως είχαμε σκοπό να προσφέρουν χρήματα η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη-μέλη, αλλά τα κράτη-μέλη έχουν προσφέρει μόνο 217 εκατομμύρια ευρώ. Φαντάζομαι πως θα μας πούν ε, πως είναι το Ευρωπαϊκό Αναπτυξιακό Ταμείο το οποίο θα πρέπει να προσφέρει. Άρα λοιπόν με τον τρόπο αυτό προσφέρουν ε, σύμφωνα και με την ε, συνεισφορά τους εκεί, αλλά παρόλα αυτά, επαναλαμβάνω, είναι λίγα τα κονδύλια που λάβαμε μέσω διμερούς ε, χρηματοδότησης. Πάρα πολλά ε, project έχουν εντοπιστεί, έχουν συμβασιοδοτηθεί και θα ήθελα να δούμε ε, κάτι το οποίο έχετε και στο φάκελό σας, που είναι η ετήσια ε, έκθεση με τα πεπραγμένα μέχρι στιγμής και έχουμε την κυρία Μοντέση σήμερα που είναι ε, από την ε, Γενική Διεύθυνση ΔΕΦΚΟ υπεύθυνη για την Αφρική και θα μας πει δύο λόγια. Ε, ξέρετε πως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εκφράσει ανησυχίες για το πώς χρησιμοποιούνται αυτά τα χρήματα και δεύτερον πώς μπορούμε να ασκήσουμε πλήρη δικαιώματα εξέτασης. Καμιά φορά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιέστε για να ε, αναλάβει δράση στα γρήγορα και δεν είμαστε ε, πάντα ενήμεροι για τις δράσεις αυτές. Επίσης, καμιά φορά ε, λαμβάνουμε μηνιαίες εκθέσεις που δεν μας δίνουν όλες τις λεπτομέρειες για το πού έχουν δαπανηθεί με συγκεκριμένους όρους αυτά τα κονδύλια για να γνωρίζουμε τι ακριβώς γίνεται. Δηλαδή, με λαμβάνουμε τις πληροφορίες αυτές αφού έχουν ε, δαπανηθεί και θα θέλαμε αυτό να βελτιωθεί. Επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει συμφωνήσει στο Διοικητικό Συμβούλιο των Επιτευμάτων να υπάρχουν και ευρωβουλευτές. Και εδώ θα πρέπει να βρούμε ποιος θα είναι ο μηχανισμός που θα μας επιτρέψει να το κάνουμε Ξέρετε πως η πρώτη συνάντηση είναι την ε, εβδομάδα ακριβώ πριν το Στρασβούργο ε, και έχουμε και κάποιες συναντήσεις Παρασκευή. Καταλαβαίνετε λοιπόν πρέπει να, πως πρέπει να βρούμε το χρονοδιάγραμμα που θα επιτρέψει στους ευρωβουλευτές να πηγαίνουν σε αυτές τις συναντήσεις. Κυρία Μοντέση, σας δίνω το λόγο για να μας κάνετε μια επισκόπηση των όσων έχουν συμβεί μέχρι σήμερα και μετά θα ακούσουμε ερωτήσεις. Uh, Πολύ σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την ε, πρωτοβουλία που αναλάβατε να μας προσκαλέσετε. Για μας είναι μια διαρκής ικανοποίηση να ενισχύουμε αυτή την επικοινωνία μεταξύ μας και να είμαστε βέβαιοι ότι υπάρχει διαφάνεια στην ε, διαχείριση των καταπιστευμάτων μας και ε, ενημέρωση του Κοινοβουλίου. Ήμουν εδώ τον περασμένο Ιούνιο για την παρουσίαση στο Κοινοβούλιο και εντωμεταξύ όπως, είπε και, όπως είπατε και εσείς πρόεδρε, έχουμε διανύμει την ετήσια έκθεση του 2016 και θα προσπαθήσουμε από το Γενάρη να υλοποιήσουμε την έκθεσή μας για το επίπεδο εκτέλεσης του 2017. Η παρουσίασή μου πρέπει να είναι σύντομη, οπότε δεν θα είμαι διεξοδική, αλλά το όντι στην έκθεση για να απαντήσω και στην ερώτησή σας, Πρόεδρε, ως προς το περιεχόμενο των όσων προσπαθούμε να κάνουμε και την προσφορά συγκεκριμένων παραδειγμάτων, εκπονήσαμε την έκθεση αυτή, δίνοντας έμφαση μέσω πινάκων στους στόχους των καταπιστευμάτων και την υλοποίηση επιτόπιων προγραμμάτων που χρηματοδοτήθηκαν. Παρόλο λοιπόν που η παρουσίασή μου δεν θα είναι τόσο διεξοδική, σας προσκαλώ να αναγνώσετε αυτή την έκθεση. Η πρόθεσή μας ήταν να παρουσιάσουμε, δεν θα παρουσιάσω τώρα τους μεγάλους στόχους του καταπιστεύματος διότι ήδη είναι γνωστοί, οι τίτλοι που σωστά θυμήσατε ε, αναφέρονται στον ίδιο το χαρακτήρα, τη φύση του καταπιστεύματος ε, του ταμείου αυτού που είναι ε, η σταθεροποίηση των χωρών του Σαχέλ, νοτιού της Σαχάρας, ε, ζώνες κρίσιμες από την άποψη της φτώχειας και των επιπέδων της, και σκοπός είναι να καταπολεμηθούν τα γενεσιοργά αίτια της μετανάστευσης, της ε, άτυπης μετανάστευσης, και κάτι άλλο που αναφέρεται επίσης στους τίτλου, η υποστήριξη των εκτοπισμένων στι ζώνες που καλύπτονται από τα καταπιστεύματα. Ο αριθμός των ε, όσων προσφέρουν χρηματοδότηση και η προστασία των εκτοπισμένων. Οι διαφάνειες παρουσιάζουν κάποιους αριθμούς από την παρουσίασή μου την τελευταία τον Ιανουάριο και το επίπεδο των ποσών που είναι διαθέσιμα. Τη στιγμή της δημιουργίας του καταπιστεύματος είχαμε ξεκινήσει με ένα ποσό 1,8 δις. Εν τω μεταξύ υπήρξαν αυξήσεις για διαφορετικούς λόγους που σας είχαμε αναφέρει στο Κοινοβούλιο και σήμερα έχουμε ένα συνολικό ποσό 2,9 δις, σχεδόν 3 δις. Εάν δούμε τους αριθμούς από την άποψη της εκτέλεσης, μπορούμε να πούμε σήμερα ότι ήδη έχουμε υποστηρίξει και χρηματοδοτήσει 117 προγράμματα για ένα συνολικό ποσό 1,9 δις, τα οποία έχουν εγκριθεί στα τρία, ε, στις τρεις τυρίδες. Για να λάβουμε υπόψη τι γεωγραφικέ ιδιαιτερότητε, τα καταπιστεύματα αποτελούνται από τρει θηρίδε μόνο. Μία για το Τσάτ και το Σαχέλ, μία για το κέρα τη Αφρική και μία για τι χώρες βορείω της Σαχάρα. 117 λοιπόν προγράμματα ήδη εγκρίθηκαν. Σε σχέση με τον στόχο που ήταν να δημιουργηθεί ένα καταπίστευμα που επιτρέπει να δράσουμε και να χρηματοδοτήσουμε γρήγορα προγράμματα. Νομίζω ότι ήδη αποδείξαμε ότι έχουμε πετύχει να ε, ε, υπάρξει επιτάχυνση σε όλε τι διαδικασίε υλοποίηση προγραμμάτων. 117 είναι αυτά που σήμερα έχουν εγκριθεί, με 169 συμβάσει να έχουν ήδη υπογραφεί. Εάν δούμε την υλοποίηση μεταξύ της έγκρισης των προγραμμάτων και της εκτέλεσής τους, έχουμε κάνει προσπάθεια επιτάχυνσης για όλη τη διαδικασία υλοποίησης των εγκεκριμένων προγραμμάτων. Από τα 117, ήδη όπως σας είπα, 169 συμβάσεις αξίας 1,2 δις. Οι αριθμοί λοιπόν στην εκτέλεση είναι ήδη ε, αυξημένοι το Κοινοβούλιο ζήτησε να ε, εντατικοποιηθούν και οι εκταμιεύσεις και αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε τους τελευταίους μήνες. Και αυτή τη στιγμή έχουμε 411 εκατομμύρια που έχουν ήδη καταβληθεί. Αυτό πραγματικά έχει να κάνει με την χειροπιαστή υλοποίηση των προγραμμάτων. Στο επίπεδο της προόδου που έχει επιτευχθεί από την προηγουμένη μας παρουσίαση, Έχουμε 23 χώρες επιλέξιμες ε, στην αρχή της διαδικασίας και σήμερα έχουμε προσθέσει άλλες τρεις. Την Κάνα, την Ακτή του Ελαφαντοστού και την Γουινέα, Κόνακρη. Ε, η διεύρυνση της ζώνης που καλύπτουμε είχε να κάνει με τη διαπίστωση, αν δούμε τις μεταναστευτικές ροές, ότι ο αριθμός των ε, υπηκόων της χώρας αυτής, Γουινεακόνα, Κρεγκάνα, Ακτήτου, Αλαφαντοστού, έχει αυξηθεί πολύ. Έπρεπε λοιπόν να υποστηριχθούν και οι τρεις αυτές χώρες στην υλοποίηση της πολιτικής μετανάστευσης για την διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε τρεις επιπλέον χώρες σε σχέση με όσα είχαμε αρχικά προβλέψει. Κυρία Πρόεδρε, αναφέρατε την κάλυψη των κονδυλίων από το καταπίστευμα. Αν δούμε το συνολικό ποσό των 2,9 δι, ε, διαπιστώνουμε ότι 2,2 δι, 2,3 περίπου, προέρχονται από το ΦΕΔ. Το μεγαλύτερο μέρος των ποσών προέρχονται λοιπόν από κονδύλια που είχαν να κάνουν με τα εθνικά ενδεικτικά προγράμματα ή τα περιφερειακά ενδεικτικά προγράμματα ή τουλάχιστον από το αποθεματικό Οπότε τα περισσότερα κάτι μέλη έρχονται και μας λένε εν τέλει την συνεισφορά μας την έχετε ήδη είναι η συνεισφορά που υπήρχε και στο ΦΕΔ και χρησιμοποιείται για αυτό το καταπίστευμα. Όμω, ήθελα να σα επιστήσω την προσοχή στο γεγονό ότι η διμερή συνεισφορά των κρατών μελών έχει αυξηθεί ιδιαίτερω. Τη στιγμή τη δημιουργία του καταπιστεύματο είχαμε όλη αυτή την απογοήτευση που και εσεί αναφέρατε, διότι υπήρχε το θέμα των συνεισφορών των κρατών ε, μελών με 83 εκατομμύρια. Όμω, ε, η δημιουργία του καταπιστεύματο επέτρεψε να αυξηθεί το ποσό. 123 εκατομμύρια επιπλέον από τα κρατημένα μελη και σήμερα έχουμε φτάσει τα 217 εκατομμύρια. Εάν κοιτάξει κανείς τις ε, συνεισφορές αυτές από την Ιταλία, τη Γερμανία και τις κάτω χώρες που έρχονται κατά κύριο λόγο, στις διαφάνειες που ε, το ε, παραδέχομαι και εγώ είναι τελείως δύσκολες, παρόλα αυτά, αν τι μελετήσετε, βλέπετε τι επιμέρου συνεισφορέ των διαφόρων κρατών μελών. Και όχι μόνο των κρατών μελών, διότι, όπω υπενθυμίστηκε σωστά, η Νορβηγία και η Ελβετία συνεισφέρουν στο κατάπιστευμα. Μία σύντομη για τη χρήση. Ποιοι είναι οι εταίροι. Ποιοι είναι αυτοί που μας βοηθούν στην ε, εκτέλεση των προγραμμάτων του καταπιστεύματος. Εάν δούμε σε αυτόν τον κύκλο τι συμβαίνει, είναι ένα ρολόι ένα κύκλος που δείχνει ότι το 47% των κονδυλίων εκτελούνται από τους οργανισμούς, τι αρχές που βρίσκονται επιτόπου από τα κράτη-μέλη. Θέλαμε δηλαδή ένα νέο εργαλείο μέσω του καταπιστεύματο που να επιτρέπει στους φορείς των κρατών μελών να συμμετάσχουν με τρόπο ε, αποτελεσματικό στην βοήθεια, την υποστήριξη της ανάπτυξης και την ε, αλληλοδιασύνδεση των προσπαθειών των κρατών μελών μεταξύ τους οι οποίες χρηματοδοτούνται εν τέλει όλες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 21% των δονδυλίων ε, εκτελούνται από τις, ανθρωπιστικές, από τις ανθρωπιστικές οργανώσεις, από τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις και επίσης υπάρχουν και διεθνείς φορείς ε, του ΟΗΕ, καθώς και ένα κομμάτι που αντιστοιχεί στους λοιπούς. Εδώ βλέπουμε λοιπόν να είναι σημαντική και η παρέμβαση του Οργανισμού για τη Μετανάστευση ή της ΥΠΑ της Αυτά ως προς την κατανομή. Θα έλεγα, εάν δείτε κατά λεπτός τους πίνακες που περιλαμβάνει η έκθεση, θα διαπιστώσετε ότι στο επίπεδο εκτέλεσης τα προγράμματα κατανέμονται με τρόπο balanced, ισόρροπο μεταξύ των διαφορών στόχων του καταπιστεύματος. Από τους στόχους κλειδιά του καταπιστεύματος έχουμε τη δημιουργία λόγου χάρη των οικονομικών ευκαιριών και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Κάτι που είναι μέρος των στόχων για την καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης ή η ενίσχυση της ανθεκτικότητας. Ανθεκτικότητα των ε, περιοχών από όπου κυρίως προέρχονται οι μετανάστες. Ή η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Ή η ενίσχυση της τοπικής διακυβέρνησης και πρόληψης των ε, συγκρούσεων. Εάν δείτε τον πίνακα ε, στο τέλος της διαφάνειας, είναι στη σελίδα 13 ή στη σελίδα 14 αυτό που σας λέω στην ετήσια έκθεση. Θα δείτε λοιπόν πως το σύνολο των χρηματοδοτήσεων κατανέμονται σωστά στους, μεταξύ των διαφόρων στόχων. Είτε πρόκειται για τους ίδιους στόχους του καταπιστεύματος, είτε για στόχους που είναι παρόμοιοι. Στόχοι που βρίσκονται και στους πέντε πυλώνες της Βαλέτας. Καλύπτονται όλοι αυτοί οι στόχοι λοιπόν. Ο στόχος αυτής της σελίδας για την παρουσίαση είναι να δώσει έμφαση ότι ένα πρόγραμμα κυρίως, οι πρακτικές δράσεις, έχει ήδη χρηματοδοτηθεί. Γι' αυτό σε αυτές τις διαφάνειες ε, βλέπετε ε, κάποια πράγματα μεμονωμένα. Έχω προσπαθήσει δηλαδή να τονίσω ότι κάποια πράγματα ήδη εκτελούνται με επίτευξη αποτελεσμάτων που σύντομα θα ε, απαριθμηθούν. Ένα πρόγραμμα που χρηματοδοτήθηκε στη Σενεγάλη λόγω χάρη για τη δημιουργία θέσεων απασχόληση. 22 θέσεις, ε, χιλιάδες θέσεις απασχόλησης δημιουργήθηκαν και επίσης για την επαγγελματική κατάρτιση με 20.000 δικαιούχους, 20.000 άτομα. Επίσης, η διάθεση τεχνικής βοήθειας για να δημιουργηθεί, δημιουργηθούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις εκεί είναι ένα παράδειγμα ένα είδος προγράμματος που καλύπτει τον πρώτο άξονα, τον πρώτο πυλώνα τέλο πάντων, δηλαδή εκτέλεση προγραμμάτων που μπορεί να διευκολύνουν τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης ή να ενισχύσουν την επαγγελματική κατάρτιση που ε, κατ' επέκταση ε, ευνοούν την πρόσβαση στην απασχόληση. Προγράμματα που ήδη λειτουργούν λοιπόν. Δεύτερο παράδειγμα, ένα πρόγραμμα στον Ήγηρα το Αζεσέν. Με αυτό προσπαθήσαμε να καλύψουμε όλους τους στόχους του πυλώνα. Στήριξη των βασικών υπηρεσιών για τον τοπικό πληθυσμό ή στήριξη της επαγγελματικής κατάρτισης. Από τη μια για τους θεσμικούς υπαλλήλους και από την άλλη για τις δυνάμεις ασφαλείας. Για τον Ιγυρά. Θέλαμε κυρίως να παρέμβουμε στο βορρά της χώρας, όπου είναι η περιοχή όπου εξοχήν υπάρχει κίνηση λαθρομεταναστών, εμπορίας ανθρώπων, και γύρω από την πρωτεύουσα, όπου προσπαθήσαμε να ε, έχουμε διαφορετικά προγράμματα ταυτόχρονα, δημιουργία θέσεων απασχόληση, στήριξη βασικών υπηρεσιών για τον τοπικό πληθυσμό και μια στρατηγική προσπάθεια ενημέρωση και ε, εκπαίδευση μάλλον και υποστήριξη των ε, διοκτικών δυνάμεων που καταπολεμούν τη λαθρομετανάστευση. 1.300 άτομα θα λάβουν εκπαίδευση σε αυτό το τομέα. Μετά αναφέρουμε τα προγράμματα IUN. Τα προγράμματα IUN, όπως ξέρετε, στόχο έχουν να δημιουργήσουν παγκόσμια εταιρική σχέση για να καλύψουμε με μια αξία μάλλον 100 εκατομμυρίων ευρώ. Και καλύπτονται διάφορες χώρες σε αυτή τη γεωγραφική ζώνη. Ήδη έχουν γίνει κάποια πράγματα, δεν θα σας δώσω τα συνολικά ποσά τώρα των μελλοντικών δικαιούχων, όταν θα έχει εξαντληθεί η εκτέλεση των συνολικών ποσών, να σας πω ότι έχει γίνει ήδη. 2.100 μετανάστες λάθρομετανάστες που έχουν μπλοκαριστεί στις μεταναστευτικές οδούς σε συνθήκες εξαθλίωσης, έχουν υποστηριχθεί, έχουν λάβει βοήθεια για να επιστρέψουν στις χώρες τους. Και έχουμε δημιουργία κέντρων IUM, τα οποία δημιουργούνται για να βελτιώσουν την εκπαίδευση, την ενημέρωση για τη μετανάστευση, τους κινδύνους από τη μετανάστευση, και να μας βοηθήσουν να συλλέξουμε δεδομένα και αριθμητικά στοιχεία που μας λείπουν ε, σε απελπιστικό βαθμό. Δεν θα σας ε, παρουσιάσω τώρα λεπτομερώς όλα τα προγράμματα, όλα τα στοιχεία περιλαμβάνονται στην έκθεση και στις διαφάνειες, αλλά προσφέρθηκε υποστήριξη στο κέρας της Αφρικής κυρίως, σε εκείνες τις χώρες, σε εκτοπισμένους ο αριθμός εκτοπισμένων είναι πολύ μεγάλος. Είναι ένα από τα βασικά προβλήματα της περιοχής, του κέρατος. Και ένα παράδειγμα η Ουγκάντα. Εκεί υποστηρίξαμε φοιτητέ και 2.100 παιδιά που είχαν εγκαταλείψει το σχολείο εκ των οποίων το 30% είναι παιδιά που προέρχονται από ε, κοινότητες εκτοπισμένων. ή μάλλον από τι κοινότητε του τοπικού πληθυσμού που ήδη βρισκόταν εκεί. Δηλαδή, μέσω τη υποστήριξη των εκτοπισμένων, καταλήγουμε να υποστηρίξουμε και τον πληθυσμό που εξασφαλίζει την υποδοχή των εκτοπισμένων. Υποστήριξη παιδιών λοιπόν της Ουγκάντας για να επιστρέψουν στο σχολείο, κάτι που κατ' επέκταση ε, εξυπηρετεί και τους εκτοπισμένους και κάτι που λόγω χάρη έγινε στη Σομαλία, όπου υπάρχει μια συνολική προσέγγιση, υποστήριξη σε παιδιά εκτοπισμένων 7.100 παιδιά υποστηρίχθηκαν και 450 άτομα έλαβαν βοήθεια για να επιστρέψουν στη χώρα προέλευσής τους. Επίσης υποστήριξε στην έναρξη μιας ενδεχόμενης οικονομικής δραστηριότητας για τα άτομα αυτά που επέστρεψαν. Στα συγκεκριμένα παραδείγματα δεν μπορώ παρά να φέρω και τα προγράμματα IUM στην Λιβύη. Στη Λιβύη, όπως γνωρίζετε, η κατάσταση είναι δραματική. Με κέντρα, με μεγάλο ρυθμό εκτοπισμένων, με μετανάστες μπλοκαρισμένους καθοδόν στις μεταναστευτικές ε, οδούς, σε συνθήκες εξαθλίωσης, σοβαρότατης. Η δράση μας στη Λιβύη σκοπό έχει να ανακτήσουμε τα άτομα αυτά, να τα βοηθήσουμε οικειοφελώς να επιστρέψουν στις χώρες προέλευσής τους. Ε, έτσι λοιπόν, τα ε, προγράμματα IUM βοήθησαν χίλιους μετανάστες που κατά την επιστροφή τους στη χώρα προέλευσης επιτυγχάνουν τους στόχους μας. Αν δούμε τους συνολικούς αριθμούς των τελευταίου εξαμήνου, μπορούμε να πούμε ότι το καταπίστευμα βοήθησε την επιστροφή και την επανένταξη 6.700 ε, λαθρομεταναστών, παράκτρομεταναστών που ήρθαν ε, ή προέρχονταν από τον ε, Νίγηρα. Στη, επέστρεψαν στη χώρα προέλευσή του. Ιδού κάποια παραδείγματα, ανέφερα μόνο μερικά προγράμματα που αφορούσαν του εκτοπισμένου, επιστροφέ μεταναστών και κάποια προγράμματα για τη δημιουργία και την έναρξη οικονομική δραστηριότητα. Δεν μπορώ όμω παρά να είμαι ε, ανακεφαλαιωτική. Στην έκθεση θα βρείτε περισσότερες λεπτομερείς πληροφορίες για τα προγράμματα αυτά. Στην έκθεση και στον ιστότοπό μας ε, εννοείται ε, υπάρχουν ακόμη περισσότερα στοιχεία. Θα ήθελα στην παρουσίασή μου επίσης να υπογραμμίσω κάτι άλλο που είναι σημαντικό και το οποίο ζητήθηκε επιμόνως και από το Κοινοβούλιο και από τα κράτη-μέλη, πώς δηλαδή φροντίζουμε για την καλύτερη δυνατή διαχείριση των κονδυλίων και πώς στην επιλογή των προγραμμάτων βασιζόμαστε στο κεντρικό χαρακτηριστικό που βρίσκεται και σε αυτή τη διαφάνεια για να παρουσιάσουμε και να στηρίξουμε τις πρωτοβουλίες μας και τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων σε στοιχεία αξιόπιστα, evidence-based που να βασίζονται στην πραγματικότητα και να προσανατολίζονται στην επίτευξη αποτελεσμάτων. Έχουμε κάνει μεγάλες προσπάθειες από την δημιουργία του καταπιστεύματος για να βελτιώσουμε αυτή τη διάσταση και αυτός ο κύκλος δείχνει πώς οι δράσεις αναλήφθηκαν σε διάφορους τομείς. Είτε σε αυτόν της έρευνας, της παρακολούθησης, της υποβολής εκθέσεων, της ανταλλαγής, της ανάληψης ε, της ευθύνης από τους δικαιούχους στα προγράμματα και την προβολή. Διαφάνεια και προβολή. Αν σταθώ στο πρώτο τμήμα του κύκλου για την έρευνα, θα πρέπει να αναφέρω ότι από τη δημιουργία του καταπιστεύματος, στα τέσσερα από τα τρία, στις τέσσερα από τις τρεις θηρίδες, δημιουργήσαμε διευκολύνσεις για την έρευνα παρουσίαση όσων έχουν γίνει εν είδη παραδείγματος για τη φυρίδα του κέρατος. Το 2016 εντοπίσαμε ένα ερευνητικό πρόγραμμα που υλοποιείται από τη Σχολή ε, Σπουδών Μέσης Ανατολής και Αφρικής του Λονδίνου όπου ζητήθηκε μια σειρά από μελέτες, αναλύσεις των γράφων εργασίας, οι οποίες να μπορούν να δυναμηθούν σε όσο το δυνατόν περισσότερου ερευνητέ, ώστε να μπορέσουμε τη στιγμή του εντοπισμού νέων προγραμμάτων να βασιστούμε σε συγκεκριμένα χειροπιαστά στοιχεία που να προέρχονται από τι ε, ερευνητικέ αυτέ μελέτε. Τα έγγραφα αυτά, οι μελέτες αυτές που είναι πιο λεπτομερείς, μας επιτρέπουν να ενισχύσουμε τον διάλογο. Διάλογο με τις δικαιούχους χώρες στα πλαίσια της διαδικασίας του χαρτούμ λόγου χάρη και σε συνεργασία με τις χώρες εταίρους. Πρόκειται για μια διευκόλυνση, ένα εργαλείο που αφορά το κέρας, αλλά παρόμοια εργαλεία έγινε, δημιουργήθηκαν και για τις χώρες του Σαχέλ. Εάν Παρό το δεύτερο σημαντικό τμήμα του κύκλου ήταν η διάσταση της παρακολούθησης κατόπιν αιτήματος και του Κοινοβουλίου, αλλά είναι και δικό μας αίτημα να παρακολουθούμε εκ του την εκτέλεση και την υλοποίηση των προγραμμάτων. Σήμερα θέλω να σας δείξω και αυτά αφορά τις τρεις θηρίδες πώς δημιουργήσαμε μια κοινή πλατφόρμα που ονομάζεται ACVO. Ένα ε, σε πραγματικό χρόνο σύστημα παρακολούθησης ένα σε πραγματικό χρονό σύστημα παρακολούθηση, το οποίο υλοποιείται απευθεία από του συμμετέχοντε στο πρόγραμμα. Είναι ένα εργαλείο δυναμικό, ευέλικτο, ε, αμήλικτο που μας επιτρέπει διαρκώς να γνωρίζουμε τι συμβαίνει με το κάθε πρόγραμμα και σε τι φάση υλοποίηση είναι. Στον ιστότοπο μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες, βλέπετε τη διεύθυνση. Επίσης, κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια για να βελτιώσουμε τη διαφάνεια και την προβολή. απευθυνόμενοι σε όλους τους πολίτες για τις διάφορες δράσεις του καταπιστεύματος. Βλέπετε εδώ την ετήσια έκθεση, που είναι ένα εργαλείο ήδη, στη σελίδα DEVCO της Επιτροπής Υπάρχει ε, συγκεκριμένη σελίδα για το καταπίστευμα. Αναγνωρίζω ότι δυστυχώ είναι περιορισμένη η σελίδα αυτή, δεν πληροφορεί τόσο γρήγορα όσο θα θέλαμε, αλλά θα δημιουργήσουμε ένα νέο ιστότοπο, ο οποίος θα απευθύνεται εντελώς και εξ ολοκλήρου ε, σε όσους ενδιαφέρονται για το καταπίστευμα. Θα είναι έτοιμος τον Οκτώβριο. Σε αυτόν τον ιστότοπο Προσπαθούμε να εντοπίσουμε γρήγορα τις πληροφορίες και τους βασικούς δρόντες, τους βασικούς φορείς, την εκτέλεση και την οργάνωση στις διάφορες χώρες και γεωγραφικές περιοχές. Και ε, εντοπίζονται και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Υπάρχει δηλαδή μια προσέγγιση στοχευμένη στα αποτελέσματα για την ε, δημιουργία αυτού του ιστοτόπου. Αυτά είναι τα εργαλεία για την βελτίωση όσων έχουν να κάνουν με τη βασική πληροφόρηση, την έρευνα, την παρακολούθηση και τη βελτίωση της επικοινωνίας μας. Κατόπιν αιτήματος της Προέδρου, μια γρήγορη ματιά στις προοπτικές για το μέλλον του καταπιστεύματος. Είδαμε προηγουμένως τα ποσά, 2,9 δις, και ήδη στην εκτέλεση έχουμε ε, εντοπίσει 1,9 δις και 800 εκατομμύρια είναι διαθέσιμα. Ποσά που είναι αρκετά περιορισμένα σε σχέση με όλες τις αιτήσει που έχουμε από τα κάτι μέλη και τις ε, συνεργαζόμενες χώρες και από τους διάφορους φορείς στην εκτέλεση που είναι διεθνείς οργανισμοί και άλλοι. Οπότε ναι, είναι σαφές ότι στο Διοικητικό Συμβούλιο τον περασμένο Ιούνιο παρουσιάσαμε άξονες προτεραιότητες για τη δράση μας. Άξονες που θα πρέπει να μας καθοδηγήσουν στην επιλογή μελλοντικών προγραμμάτων που θα χρηματοδοτηθούν φέτος και το 2018. Οι διαφάνειες αυτές ε, αναφέρουν κάπως αυτούς τους άξονες, τις στρατηγικές προτεραιότητες. Εάν δεν κανείς τις στρατηγικές προτεραιότητες που αναφέρονται γεωγραφική ζώνη, γιατί για άλλη μια φορά οι προτεραιότητε και η κατάσταση στις διάφορες περιοχές διαφέρει και μας οδηγεί να κάνουμε επιλογές που δεν είναι όλες ίδιες, αλλά είναι συνεχείς μεταξύ τους, ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε περιοχής. Ας πάρουμε το κέρας. Στο κέρας θα πρέπει να συνεχίσουμε να στηρίζουμε προγράμματα για την υποδοχή μεταναστών. Είναι μια περιοχή με 3 εκατομμύρια, πάνω από 3 εκατομμύρια μετανάστες και εκτοπισμένους, το μεγαλύτερο αριθμό εκτοπισμένων και μεταναστών τον εντοπίζουμε ακριβώς εκεί, στο Κέρας. Οπότε θα πρέπει να συνεχίσουμε να στηρίζουμε αυτά τα διάφορα προγράμματα. Επίσης υπάρχουν δράσεις στον τομέα της καταπολέμησης της ε, εμπορίας για να εντοπίσουμε όλες τις πηγές της μετανάστευσης τις οδούς που απλώς περνούν από το κέρας για να προχωρήσουν προς την Ευρώπη. Σε ό,τι αφορά το Σαχέλ και το Τσάντ και εκεί προτεραιότητα στις μελλοντικέ μας δράσεις θα είναι κάποια θέματα κλειδιά. Ένα, η καταπολέμηση και ενίσχυση του διαλόγου για τη μετανάστευση. Όπω γνωρίζετε, για την κάθε χώρα έχουμε θεσπίσει εταιρικέ σχέσει για τον διάλογο περί μετανάστευση, διάλογο που τον παρακολουθούμε με δράσεις καλής διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών. Για να ε, ευνοήσουμε και την επιστροφή και επανένταξη. Δεύτερη διάσταση, σταθεροποίηση. Στην περιοχή του Σαχέλ στη γεωγραφική ζώνη που μας φέρνει πιο κοντά στις πηγές της λαθρομετανάστευσης. Υπάρχουν περιοχές που είναι τελείως αποσταθεροποιημένες, εγκαταλελειμμένες από τα κράτη τους. Περιοχές όπου εγκαθίστανται εύκολα όλοι οι εξτρεμιστές και οι εξτρεμιστικές δυνάμεις. Πρόκειται για περιοχές που θέλουμε να τις στηρίξουμε με ανάπτυξη με δράσεις για να διευκολύνουμε την προσφορά βασικών υπηρεσιών, με δράσεις για να ενισχύσουμε το επίπεδο ασφάλειας και την ε, δράση των ιδιωτικών δυνάμεων. Τρίτη διάσταση, τρίτη φυρίδα για την Βόρεια Αφρική. Θα έλεγα ότι ο όγκος, το ποσό των κονδυλίων που διατίθενται θα επικεντρωθούν στην μετανάστευση και την ε, παράτυπη μετανάστευση για άλλη μια φορά για να συνεχίσουμε να προσφέρουμε την απαραίτητη βοήθεια, την πληροφόρηση, να διευκολύνουμε την επανένταξη των εκτοπισμένων και των παράτυπων μεταναστών που βρίσκονται σε αυτή τη μεταναστευτική οδό, αλλά και με δράσεις που θα διευκολύνουν, θα έλεγα, την νόμιμη μετανάστευση και την κινητικότητα για αυτές τις χώρες που είναι κλειδί για την καλή συνεργασία με όλε τι χώρε εταίρου. Ιδού οι τρει προτεραιότητε, θα έλεγα οι άξονα προτεραιότητα στρατηγική δράση που έχουμε παρουσιάσει και στο Διοικητικό Συμβούλιο. Πράγματι, με αυτούς τους τρεις άξονε δράση. το συμπέρασμα είναι ότι θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να συνεχίσουμε να εκτελούμε δράσεις με μεγαλύτερη προτεραιότητα στις διασυνοριακές δράσεις, στις διαθυριδικές δράσεις και σε όσες θα μας επιτρέψουν να αντιμετωπίσουμε προκλήσεις που σήμερα είναι μεγάλων διστάσεων. Τα είδατε και στον τύπο. Αναφέρθηκε η πρωτοβουλία των Βερσαλιών μετά τις συζητήσεις στο Παρίσι. Πρωτοβουλίες για να συγκεντρώσουμε το σύνολο δράσεων και να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση τόσο στο βόρειο, στη Βόρεια Αφρική, όσο και στις υπόλοιπες χώρες ε, νοτίως της Σαχάρας. Θα πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε να επιδιώκουμε μια προσέγγιση balanced, μια ισόρροπη προσέγγιση μεταξύ διαφόρων δράσεων και στόχων όπως αναφέρθηκαν στη Βαλέτα. Οι προτεραιότητες αυτές είναι προτεραιότητες για τις συγκεκριμένες μας δράσεις όπως ορίστηκαν στο πλαίσιο του Συμβουλίου. Συμπεράσματα τα οποία ε, απεστάλησαν και στο Κοινοβούλιο, τα οποία μπορείτε να δείτε λοιπόν, και αναφέρθηκαν και σε αυτή την παρουσίαση. Αυτά. Ίσως θα πρέπει να πάψω εδώ. Ελπίζω ότι αξιοποίησα στο μέγιστο βαθμό τη χρόνο που μου διατέθηκε, αλλά θέλω να υπάρξει χρόνος και για να απαντήσω στις ερωτήσεις σας η υπεύθυνη διαχείριση του καταπιστεύματο, τι διάφορε θηρίδε του καταπιστεύματο, είναι εδώ μαζί μου στην αίθουσα. Με μεγάλη χαρά θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στο σύνολο των απορριών σας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ και χαίρομαι που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε ε, μια αρκετά εκτενή τέτοια παρουσίαση γιατί βλέπουμε ότι οι συνάδελφοι προφανώ ενδιαφέρονται πάρα πολύ το θέμα αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα. Το, ο κόσμο θέλει να το κατανοήσει, θέλει να κατανοήσει σε βάθο το θέμα τη ε, μετανάστευση στη Μεσόγειο. Αποτελεί ασφαλώ και θέμα πολιτική προτεραιότητα. Πάρα πολλοί συνάδελφοι λοιπόν έχουν ζητήσει τον λόγο. Ένας από κάθε ομάδα και μετά θα έχουμε κι άλλον ένα γύρο. Ο κύριος Πρέντα πρώτος. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την παρουσίαση. κύριε Μοντάζη. Μία παρατηρήση, επιτρέψτε μου καταρχάς, γενικής φύσεως. Και στη συνέχεια θα ήθελα να σας θέσω και δύο ερωτήσεις. Η γενική παρατηρήση είναι η εξής. Για τα τρία τις τρεις θηρίδες τις οποίες αναφέρατε, Τσάτ, ε, το κέρας της Αφρικής και η Βόρειος Αφρική. Είδα την κατανομή των πόρων 40, 40 και 20% αντιστοίχως για τις τρεις αυτές θηρίδες. Η παρατήρηση την οποία θα ήθελα να κάνω είναι η εξή. Ενδεχομένω και να πρέπει να αναλογιστούμε συντόμως το πώς θα εξισορροπηθούν αυτές οι τρεις θηρίδες, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το, τη θηρίδα που αφορά τις χώρες της Βορειάς Αφρικής, Αλγερία, Μαρόκο, την Ισία και η Αίγυπτος, η οποία προστίθεται στις χώρες του Μαγκρέπ το καινούριο στοιχείο είναι ότι οι χώρες αυτές δεν είναι μόνο χώρες προέλευσης μεταναστών, όλο και πιο πολύ γίνονται και χώρες διέλευσης μεταναστών, μεταναστών που προέρχονται από το Σαχέλ. Πρόκειται και για χώρες δε που αποτελούν και προορισμό των μεταναστών όπως το Μαρόκο, η Αλγερία και η Τινησία. Με διαφορετική αντίδραση κάθε φορά των αρχών των χωρών αυτών. Ε, οι Μαροκινοί, για παράδειγμα, δίνουν χαρτιά σε μεγάλο ρυθμό τέτοιων μεταναστών από την ε, υποσαχάριο περίοδο. Η Αλγερία όλο το θερινό διάλειμμα συζήτησε επισταμένως ε, τι θα γίνει με τους μετανάστες, κατά πόσον θα δίνεται άδεια. Και υπήρχε και το θέμα της απαγόρευσης και στην Τινησία διεξάγα για την ανάλογη συζήτηση. Οι χώρες λοιπόν αυτές ε, στη Βόρεια Αφρική δεν είναι πλέον χώρες μόνο ούτε προέλευσης ούτε διέλευσης μεταναστών αλλά και χώρες προορισμός. Στο Μαρόκο, για παράδειγμα, γίνεται συζήτηση για τα προγράμματα τα οποία υπάρχουν ήδη στο Μαρόκο για να επανέλθουν, να επιστρέψουν οι μετανάστες, αλλά φυσικά και το θέμα των νέων μεταναστών. Αυτό ως γενική παρατηρήση. Δύο ερωτήσει τώρα, επιτρέψτε μου. Η πρώτη για τη συμβολή των κρατών μελών. Αυτό που θα ήθελα να ξέρω, γιατί δεν το είδα αυτό πουθενά ως πληροφορία, δεν ξέρω το παρέβλεψα κάπου, αυτές οι συμβολές, οι συνεισφορές είναι στόχοθετημένες, για παράδειγμα, όταν οι Σλοβάκοι και οι Αυστριακοί έχουν πόρους να συνεισφέρουν. Λένε για παράδειγμα ότι αυτοί οι πόροι θέλουμε να πάνε στο Τζιμπουτί, θέλουμε να πάνε στο Τσάτ ή απλά έτσι γενικά δίνουμε κονδύλια γενικά σε οργανώσεις ε, οι οποίες με τη σειρά τους κάνουν, ε, αν θέλετε, την ε, στόχοθέτηση. δεύτερη ερώτηση σε ό,τι αφορά την προσανατολισμό των έργων, σε ό,τι αφορά τις ΜΚΟ και που αποτελούν και τους πιο δραστηριοποιημένους, αν θέλετε, φορείς βλέπω και τα σχετικά ποσοστά σε ό,τι αφορά τις ΜΚΟ. Οι ΜΚΟ λοιπόν αυτές είναι τοπικές οργανώσεις ή ευρωπαϊκές. Έχετε κάπως πιο ακριβή στοιχεία να μας δώσετε σε ό,τι αφορά τους ε, διεθνείς φορείς που δραστηριοποιούνται σε σχέση και με τους τοπικούς φορείς δηλαδή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ λοιπόν για την παρουσίασή σας και είμαι πεπισμένος ότι θα μας δώσετε ικανοποιητικές απαντήσεις. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ αλλά και πρόεδρος, ο κύριος Νόιζερ, ο Νόρμπερτ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσίαση. Μία παρατηρήση έχω να κάνω για την χρηματοδότηση. Μισό λεπτό, ναι. Η δική μου παρατηρήση έχει να κάνει λοιπόν με τα θέματα χρηματοδότησης ε, του καταπιστεύματος. Όπως και σε πολλά άλλα έργα, η χρηματοδότηση είναι εντελώς ασαφής. Υπάρχουν πάρα πολλές διαφορετικές πηγές χρηματοδότησης και επί της αρχής δεν μπορούμε να ελέγξουμε τι χρήματα δίνει το κάθε κρατός μέλος. Ακούμε και το επιχείρημα ότι, α, κοιτάξτε, εμείς ήδη συνεισφέρουμε, συμμετέχουμε ήδη σε προγράμματα. Αυτό δεν το λέω ως κατηγορία, ως, ε, δεν το προσάπτω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά πιστεύω ότι είναι απαραίτητο να ξεκαθαρίσουμε πώς και σε τι βαθμό συνεισφέρουν τα κράτη-μέλη στα ταμεία αυτά. Δεύτερη ερώτηση. Σε ό,τι αφορά την διάσκεψη η οποία έλαβε χώρα στο Παρίσι, τέσσερα μεγάλη μέλη: Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία και Ιταλία. Συναντήθηκα με την Ιγυρία, το Τσάντα και τη Λιβύη, τρία μεγάλα κράτη στην Αφρική. Οι δραστηριότητε αυτές πώς αντιμετωπίζονται από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γιατί εδώ θεωρώ ότι ανεξάρτητα από αυτά που γίνονται στην Ευρωπαϊκή Αναπτυξιακή Βοήθεια, αναζητούνται συγκεκριμένες ε, λύσεις, οι οποίες όμως ε, δεν ε, στις οποίες δεν συμμετέχει ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση επαρκώς, ούτε η ειδική εντεταλμένη αυτές οι μεμονωμένες δράσεις, όσο ευγενείς και να είναι, θα έπρεπε να έχουν τις βάσεις τους στην ευρωπαϊκή διαδικασία, πιστεύω. Ο κύριος Βάβενεν και μετά η κυρία Σαρχεντίνη. Σας ευχαριστώ και θα μιλήσω φιλανδικά. Δύο ερωτήσεις έχω να κάνω. Και ο κύριος Πρέντα και ο κύριος Νόιζερ μίλησαν για το ρόλο των κρατών μελών σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση του καταπιστεύματος. Φυσικά είναι μεγάλη απαγοήτευση ότι δεν, χρησιμο, ότι δεν συμμετείχαν πιο εντατικά τα κρατη γιατί το όλο σύστημα βασιζόταν στην αρχή ότι τα κρατη θα συμμετείχαν ισότιμα στην χρηματοδότηση του καταπιστεύματος. 50% περίπου των πόρων διανέμονται μέσω των αρχών συντονισμού των κρατών μελών. Αυτό τι σημαίνει, τα κράτη-μέλη έχουν συνεισφέρει λιγότερους πόρους ό,τι αφορά την ανάπτυξη όταν ξεκίνησε ο συντονισμός των πόρων αυτών για το καταπίστευμα. Ε, πρόκειται για ένα καταπίστευμα, ξέρετε, εκτάκτου ανάγκης και τώρα φαίνεται ότι εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ έχουν ήδη χορηγηθεί. Δεν μπορεί να γίνει πιο ταχεία αυτή η διαδικασία σε ό,τι αφορά το καταπίστευμα. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ και έχουμε πολλά συγκεκριμένα ερωτήματα, λέει η Πρόεδρο, η κυρία Σαρχεντίνη. Και μετά θα σταματήσουμε να ακούσουμε τι απαντήσει και μετά θα ακολουθήσει η δεύτερο γύρο, η κυρία Σαρχεντίνη. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σα ζητώ συγγνώμη, αλλά νομίζω ότι ακόμα δεν έχουμε πετύχει σωστό έλεγχο για το καταπίστευμα. Ακόμα αγωνιζόμαστε. Βλέπουμε την ετήσια έκθεση του 2016. Ε, το όλοι την έχουμε δει. Δεν αποτελεί αυτό όμως εποπτεία. Σωστή. Έχει περάσει και πολύ καιρό. Σεπτέμβριο έχουμε πλέον και βλέπουμε κάποια γενικά στοιχεία που μας δίνει μια γενική εικόνα και πιστεύω ότι το καταπίστευμα διαρκώς θα πρέπει να δικαιολογεί γιατί δεν ακολουθεί τις συνήθεις οδούς ανάπτυξης. Γιατί ε, επιτρέπεται να υπάρχει χαμηλότερο επίπεδο ελέγχου και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Η δικαιολογία ότι το καταπίστευμα αυτό ε, πρέπει να δραστηριοποιείται πιο γρήγορα είναι ένα συνηθισμένο επιχείρημα. Αλλά παρόλα αυτά πιστεύω ότι θα πρέπει αυτό ενδεχομένω να σημαίνει ότι θα πρέπει να, επιληφ... να επιληθούν προβλήματα στο EDF, στο DCI, αλλά όχι να αφαιρεθεί και να μειωθεί το επίπεδο ελέγχου. Για να καταλάβουμε λοιπόν ποιο είναι το αποτέλεσμα, το πραγματικό αποτέλεσμα των δράσεων αυτών, θα έπρεπε να το συγκρίνουμε δίπλα-δίπλα με τα προγράμματα που έχουμε συμφωνήσει στον DEF σε ό,τι αφορά τα εθνικά προγράμματα, τα αντικτικά προγράμματα, προκειμένου να έχουμε μια σωστή σύγκριση. Ο καθένας προσωπικά, αλλά και για την ομάδα του, για να αποφασίσουμε αν όντως αξίζει τον κόπο η μειωμένη εποπτεία. Εγώ δεν μπορώ να πω ότι μπορώ να το κάνω με τα στοιχεία που έχω στη διάθεσή μου και αυτό πιστεύω ότι αποτελεί μεγάλο πρόβλημα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Μια χώρα η οποία είναι στο καταπίστευμα για την Αφρική. Η, ακρι... η ακτή του ελεφαντοστού. Πήγαμε στο Αμπίτζαν για την διάσκευση, το εξέτασα λοιπόν τα στοιχεία αυτά και αναρωτήθηκα κατά πόσο μήπω υπάρχουν προγράμματα τα οποία θα μπορούσα να επισκεφτώ στην ακτή του ελεφαντοστού σε σχέση με το καταπίστευμα δηλαδή από το Φεβρουάριο συγκαταλέγεται στις χώρες αυτές ε, η ακτή του έλεφαντος του και από τις αναλήψεις προκύπτει ότι είναι μεγάλο το τμήμα της νεολαίας, ε, ότι μεγάλο το τμήμα της νεολαίας ε, φεύγει για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα συνηθισμένα για την ανεργία της, των νέων, για τις ευκαιρίε που πρέπει να χορηγηθούν στους νέους. Τα project τα οποία συμπεριλαμβάνονται είναι ένα πρόγραμμα για τη διαχείριση της ε, μετανάστευσης και ένα άλλο είναι ένα πρόγραμμα ενημέρωσης για την ε, δυτικοαφρικανική αστυνομία. Θα ήθελα να καταλάβω πώς αυτή η ανάλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η ακτή του ελεφαντός του σε ό,τι αφορά την ενεργεία σχετίζεται με αυτά τα δύο συγκεκριμένα προγράμματα για τη διαχείριση δηλαδή της μετανάστευσης και για την... τα συστήματα ενημέρωσης της αστυνομίας. Εγώ δεν τα βγάζω. Δεν μου βγαίνει το σύνολο το άθροισμα. Τι σχέση έχει αυτό. Θα ήθελα να καταλάβω λοιπόν κατά πόσον όλα αυτά πραγματικά εκπληρώνουν τους στόχους τους οποίους έχουμε θέσει. Δεν μπορώ να το συμπεράνω αυτό από τα στοιχεία που έχω στη διαθέσή μου. Έχουμε μία ομάδα ελέγχου και εποπτείας, ιδιαίτερα για την ε, μετανάστευση και έγινε και μία μεγάλη διάσκευση για τον Ήγηρα και θα σταματήσω το σημείο αυτό, Πρόεδρε. Αλλά αυτό που προέκυψε από τη διάσκεψη αυτή για τον Ήγηρα είναι ότι πραγματικά δαπανούνται κονδύλια και πραγματικά γίνεται ε, σωστή δουλειά για να εντοπιστούν οι διακινητές, αλλά υπάρχει και μεγάλη ανεργία την οποία εμείς την δημιουργήσαμε. Γιατί αυτός ο κόσμος έκανε φυσικά εγκληματικές δραστηριότητες, αλλά τι θα βοηθήσει αν μείνουν στο δρόμο και δεν έχουν δουλειά. Αυτό αποσταθεροποιεί ε, τον κόσμο και τίποτα δεν επιθέτει πάνω από μια κοινωνία από την ενεργεία των νέων. Δεν μπορώ να κρίνω, πέρα δηλαδή από την ανάλυση που έχουμε για το 2016, ποια είναι τα αποτελέσματα, ποιο είναι αυτό που πετύχαμε. Το έχω ξαναπεί στο παρελθόν, θεωρώ. Αλλά για να υπάρχει σωστός έλεγχος χρειαζόμαστε πολύ παραπάνω στοιχεία. Σας ευχαριστώ να ακούσουμε και τον κύριο Σαφάουζερ στο γύρο αυτό. Καλημέρα σας. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρία μου. Θα ήθελα και σε εσά να ευχηθώ καλημέρα, μια που σήμερα είναι η πρώτη μέρα της επιστροφής. Νομίζω πως η πρωτοβουλία αυτή είναι πολύ καλή. Πρώτα απ' όλα γιατί αντιμετώπισα σε όλη μου την καριέρα στα θέματα τα αναπτυξιακά ένα σωρό ταμεία με κονδύλια τα οποία ποτέ δεν εκταμιεύθηκαν. Το γεγονός λοιπόν ε, της δημιουργίας ενός καταπιστεύματος, ενός ταμείου ε, αντί των ε, διαδικασιών που συνήθως ακολουθούμε είναι πολύ θετική. Δυστυχώς έφτασα αργά, θέλω όμως κάποιες εξηγήσεις. Να σας πω πως εγώ καταρχήν είχα, ήμουν επικεφαλής ε, ενός ιδιωτικού ταμείου ε, με μια επιτροπή ε, επενδυτική στην οποία συγκεντρώνονται όλοι οι δωρητές. Εκεί τα κράτη προσφέρουν τις συνεισφορές τους και βέβαια να σας πω πως έχουμε και το κομμάτι που αντιστοιχεί ε, στα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, από τα διάφορα ταμεία, αλλά βεβαίως υπάρχει και διαχειριστική επιτροπή. Και νομίζω πως στην ε, περιοχή αυτή, και σύντομα θα ξαναπάω στο Μαλί και στην Κεντρική Αφρική και αυτό που διαπιστώνω εκεί είναι πως χρειάζεται οπωσδήποτε να στήσουμε project. Όχι δηλαδή να περιμένουμε να μας τα φέρουν για να τα χρηματοδοτήσουμε ή να τα δημιουργήσουν οι μη καπαόμικρον. Όχι. Θα πρέπει εμείς να δημιουργήσουμε project έτσι ώστε να υπάρχουν συνθήκες απασχόλησης, εργασίας, έτσι ώστε όντως να σταθεροποιήσουμε τον πληθυσμό που βρίσκεται επί τόπου και να βρούμε άλλα πτυξιακέ τοπικές λύσεις. Και γι' αυτό πιστεύω πως χρειάζεται μια ιδιωτική επιχείρηση η οποία ε, με τη μορφή της Διαχειριστικής Επιτροπής θα διαχειρίζεται όλα αυτά τα project, θα τα αναλαμβάνει. Αυτή λοιπόν η διάσταση υπάρχει ως δυνατότητα στο δικό σας καταπίστευμα. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Και η δεύτερη, εάν όχι, δεν θα έπρεπε να το κάνουμε έτσι ώστε να έχουμε ΣΔΙΠ έτσι ώστε ανάλογα με το project σε κάθε περίπτωση για μια χώρα ή για μια ζώνη, μια περιοχή χωρών να και μιλώ εδώ για την οικονομική ανάπτυξη, να δημιουργούμε project τα οποία θα φέρουν απασχόληση και βέβαια θα έχουν και κάποιο είδους απόδοση επενδυτικά. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Πολλές ερωτήσεις που ακούσαμε, πολύ συγκεκριμένες και πολύ σχετικές. Πρέπει να σας πω πως σοκαρίστηκα από την εξή είναι παρόλο που ανακυκλώνω, επειδή α, ανακυκλώνονται αυτά τα κονδύλια, έχουμε τα επιπρόσθετα αυτά, αυτό το ελέγχεται. Επίσης η ισορροπία μεταξύ περιφερειών και τα λοιπά, Νομίζω ότι ήταν συγκεκριμένες ερωτήσεις και θα δώσετε συγκεκριμένες απαντήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Να σας ευχαριστήσω για τις ερωτήσεις σας. Και καταλαβαίνω απόλυτα το ότι αισθάνεστε κάποιο ε, εκνευρισμό. Εγώ σας τα είπα στα γρήγορα και θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες για όλες τις δράσεις. Και γι' αυτό ήθελα να σας δείξω πως είναι εύκολη πρόσβαση πληροφορίε αν ξέρετε πού να ψάξετε. Αλλά για να απαντήσω σε ερωτήσεις σας, Θα ακολουθήσω τη σειρά με την οποία ακούστηκαν. Καταρχήν, κατανομή κονδυλίων. Όταν τα κονδύλια, όταν δημιουργήθηκε αυτό το καταπίστευμα, δημιουργήθηκε από πόρους που προέρχονται από διάφορα χαρτοφυλάκια. Θα πρέπει λοιπόν την νομιμότητα στη διαχείριση αυτών των ταμείων να τη Οπότε κατανείμαμε τα, τα, τα κονδύλια ανάλογα με την προέλευση αυτών των ταμείων. Και σύμφωνα με τα όσα έχετε εκεί στον Πίνεκα το μεγάλο κομμάτι αυτών των 2,3 δις προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης. Άρα λοιπόν μπορούν να διατηθούν μόνο στις χώρες που καλύπτονται από το ταμείο αυτό. Αν σε αυτό προσθέσουμε ε, τα διάφορα ταμεία που προέρχονται από, ε, κονδύλια που προέρχονται από άλλα ταμεία, από το Ταμείο Γυπνίασης, από ε, το ΝΟΙΕ, θα δούμε πώς μπορούμε να καλύψουμε και τις χώρες της Βορείου Αφρικής και να δούμε τι γίνεται με τη διαχείριση αυτών των κονδυλίων, γιατί βλέπουμε πως έχουμε πολύ περισσότερα κονδύλια που απευθύνονται στη Βόρεια Αφρική ε, γιατί η κατανομή όπως σας είπα είναι 40-40-20 βασιζόμενη στην ανάγκη που έχουν διάφορες χώρες είναι μια πολιτική απόφαση και σεβόμενη τα διάφορα χαρτοφυλάκια και ε, την, ε, τα, τους κανονισμούς των ταμείων από την οποία προέρχονται τα χρήματα αυτά. Σεβόμαστε αυτή την κατανομή, είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε, και όταν φτάνουμε σε αυτό το καταπίστευμα, ξέρετε πως πήραμε πάρα πολλά κονδύλια, πολλά κονδύλια από τα εθνικά ενδεικτικά προγράμματα, από τα περιφερειακά προγράμματα, 200 εκατομμύρια για παράδειγμα, από το περιφερειακό πρόγραμμα για την Δυτική Αφρική, τα οποία πήραμε από εκεί και τα βάλαμε στο καταπίστευμα. Άρα λοιπόν και εκεί θα πρέπει να σεβαστούμε τους κανονισμούς, γιατί έχουμε κάποια ε, χρήματα που θα έπρεπε κανονικά να πάνε απευθείαν στι χώρε της Δυτικής Αφρικής και τα μεταφέραμε στο καταπίστευμα. Άρα λοιπόν σε πολιτικό επίπεδο θα πρέπει να σεβαστούμε το ότι τα χρήματα αυτά πηγάζουν από εκεί. Όχι μόνο λοιπόν στι νομικέ διαδικασίε, αλλά και σε πολιτικό επίπεδο. Παρ' όλα αυτά καταλαβαίνω την δυναμική τη απάντησή σα, και σήμερα αν εξετάσει κανεί την διαχείριση των ροών ε, το πρόβλημα είναι η Λιβύη. Πρέπει λοιπόν να διευκολύνουμε τη χρηματοδότηση των διασυνοριακών ή διαθυριδικών προγραμμάτων για να στηρίξουμε και να συνεισφύρουμε έτσι ώστε στην θηρίδα τη μία ή την άλλη να βρούμε κονδύλια που θα μας επιτρέψουν ε, ε, την επιστροφή ατόμων που είναι μεν από χώρες της ε, Μαύρης Αφρικής αλλά έχουν περάσει από τη Λιβύη. Και όλα αυτά εξετάζοντας τι γίνεται και με την ε, επιστροφή ανθρώπων από την Ιγυρία, από τον Ήγυρα και πώς θα καταφέρουμε να επιστραφούν αν έχουν περάσει από τη Λιβύη. Αυτό είναι μια προτεραιότητα για τις επόμενες φάσεις. Και θα πρέπει έτσι να έχουμε αυτή τη θηρίδα στο βορρά ε, ε, τη θηρίδα του Βορρά χρησιμοποιώντας και την θηρίδα του Σαχέλ, όμως με συμμόρφωση και σεβασμό στις νόμιμες διαδικασίες. Για την παρουσίαση που έκανα για την κατανομή των κρατών μελών, ξέρω πως ο πίνακας αυτός είναι δυσανάγνωστος, δεν έχω PowerPoint άλλο να σας δείξω, αλλά το έχετε στην έκθεση και το βρίσκετε και στο site μας. Άρα λοιπόν μπορείτε να το δείτε οποιαδήποτε στιγμή και θα σας δείξει αυτό ποια είναι η χρηματοδότηση κράτος ανακράτος τρίτων χωρών κρατών μελών. Για παράδειγμα, τι έχει συνεισφέρει η Ελβετία, η Νορβηγία. Είναι από την ετήσια έκθεση τα στοιχεία, αλλά την έχουμε την έκθεση την ετήσια και μπορείτε να τη δείτε όποτε θέλετε. Η Ιταλία σύντομα θα αποφασίσει να συνεισφέρει κατά 2 εκατομμύρια τη συνεισφορά του, Μόλις τα λάβουμε με την επιστολή που επιβεβαιώνει αυτή τη συνεισφορά θα ενημερώσουμε αμέσως αυτόν τον κατάλογο. Ο πίνακα λοιπόν θα αλλάξει. Άρα λοιπόν οι πληροφορίε για τι συνεισφορέ των κρατών μερών ε, είναι διάφανος και βρίσκεται κάθε στιγμή στη σελίδα μας στο διαδικτύο. Τώρα, για τη συνεισφορά αυτή των κρατών μελών, ε, ε, ακούστηκε και μία ακόμα ερώτηση. Δηλαδή, στόχευση. Στόχευση. Δύο ευρωβουλευτές μου το ζήτησαν. Να σας πω πως τη στιγμή που μεταφέρουμε ε, κονδύλια ανεξάρτητα με το φάκελο και με το κράτος μέλος θα πρέπει όλα αυτά να συγχωνεύονται σε ένα ενιαίο πακέτο. Βέβαια, σε πολιτικό και στρατηγικό επίπεδο λαμβάνουμε υπόψη τις προτεραιότητες που έχουν παρουσιαστεί τη στιγμή που έχουμε ακούσει τις, ε, λάβει τις ε, διμερείς κάποιων χωρών. Δηλαδή, κάποια στιγμή έρχονται τα κράτη, μέλη και μας λένε «Κοιτάξτε, θα συνεισφέρω, αλλά θα ήθελα ε, κυρίως να πάει ε, στη Θηρίδα, Βορειοφρική, Σαχέλ κτλ. Άρα λοιπόν γίνεται μια τέτοιου είδους στόχευση και παρουν κρατη κράτη-μέλη, για παράδειγμα η Ιταλία, που έρχεται και λέει θα ήθελα οπωσδήποτε να ενισχύσω τη δράση μας στον Ήγηρα, αλλά μέσω καταπιστεύματος. Γιατί έχει κάποια πλεονεκτήματα, συνέργειες για παράδειγμα, συμπληρωματικότητα με άλλα κράτη-μέλη. Άρα λοιπόν ακούμε αυτές τις προτάσεις για τη στοχευμένη χρήση και βεβαίως ενισχύουμε το ποσό το οποίο πάει για τον Ήγυρα χρησιμοποιώντας παρόλο που δεν υπάρχει για παράδειγμα συγκεκριμένη χρήση μέσα στον πολυπλογισμό, συγκεκριμένη γραμμή μέσα στον προπολογισμό, αλλά θα το κάνουμε με τον τρόπο που μας ζήτησε η Ιταλία μέσω τη συνεισφορά τη. Το μέσο λοιπόν, έτσι ώστε για να διαχειριστούμε ε, τα κονδύλια αυτά υπάρχουν. Ξέρετε πως τα κράτη-μέλη στην αρχή ήταν ε, διστακτικά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην αρχή ήταν πολύ φιλόδοξη. Είχε πει ένα δις εμείς, ένα δις τα κράτη-μέλη. Αυτό δεν συνέβη. Αλλά το γεγονός πως η συνεισφορά αυτών των κρατών μελών όσο περνάει ο καιρός μεγαλώνει, αποδεικνύει πως αυτό το καταπίστευμα είναι επιτυχημένο και δημιουργεί πρωτοβουλίε οι οποίε είναι συμπληρωματικέ μεταξύ του και έχουν συνέργεια. Δηλαδή θα πρέπει να χρησιμοποιούμε με πιο γρήγορο τρόπο το ταμείο αυτό και νομίζω ότι το κάναμε ήδη. Ε, ε, αποδείχθηκε και γι' αυτό το χρησιμοποιούν περισσότερο τα κράτη-μέλη. Ιταλία, Γερμανία, όλη τη συνεισφορά τους ε, για το Σαχέλ και για την διαχείριση των μεταναστικών ροών τη στέλνουν μέσω καταπιστεύματο, Έτσι ώστε να προχωράμε με πολύ πιο γρήγορα βήματα. Ακούστηκε και μία ακόμα ερώτηση για την ταχύτητα εκτέλεσης και πρέπει να σας πω πως έδωσα τα στοιχεία μόλις ξεκίνησα την παρουσίασή μου. Καταλαβαίνω πως δεν είμαστε ικανοποιημένοι, αλλά αν συγκρίνουμε τα στοιχεία που έχουμε με τι γίνεται στο κανονικό Ταμείο ε, Ανάπτυξης, θα δείτε πως εμείς είμαστε πολύ πιο γρήγοροι. Βεβαίως, πετύχαμε να επιταχύνουμε όλες τις διαδικασίες έγκρισης για τα project. Είναι ξεκάθαρο πως κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να επιταχύνουμε την υπογραφή των συμβάσεων και είναι ξεκάθαρο πως επί τόπου, τη στιγμή των διαφορών δράσεων, οι εταίροι μας αντιμετωπίζουν προκλήσεις οι οποίες πραγματικά καμιά φορά είναι τεράστιες. Εντάξει, δεν είναι συνεργασία με χώρες τα οποία όλα είναι εύκολα. Μιλάμε για project τα οποία εφαρμόζουμε σε ζώνες οι οποίες είναι στην έρημο ή σε περιοχές οι οποίες δεν είναι καθόλου προσπελάσιμες για λόγους ασφάλειας. Οπότε κάναμε ό,τι μπορούμε για να επιταχύνουμε την εφαρμογή. Μιλάμε με υπηρεσίες και με θεσμούς στα κράτη-μέλη έτσι ώστε να επιταχύνουν και αυτές τα όσα κάνουν και την παρουσία τους επιτόπου. Αλλά ξέρετε πως το να είναι κανείς επιτόπου πολλές φορές αποτελεί τεράστια πρόκληση και είναι πολύ λίγη η προσπελασιμότητα σε περιοχές ε, στις οποίες έχουμε ξεκινήσει δράση με τοπικούς φορείς οι οποίοι θα πρέπει ε, να μας δεχτούν ε, και να κατανοήσουν το ποια είναι η δράση μας. Τώρα, για το τι συνέβη στο Παρίσι και την εκδήλωση εκεί. Να πω πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν πλήρως ενταγμένη και στην προετοιμασία ε, και στην εκτέλεση. Βέβαια τον ηγετικό ρόλο είχε η Γαλλία. Συγκάλεσε τη συνάντηση. Ήταν όμως εκεί όλες οι χώρες. Το περιεχόμενο της δήλωσης προετοιμάστηκε με τη συνεργασία της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και ήμασταν εκεί. Ήταν εκεί η ύπατη εκπρόσωπος, όχι μόνο όμως λόγω της, ε, του χαρτοφυλακίου της, αλλά και ως αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κυρία Μογκερίνη. Οπότε ήταν μια στρατηγική συνάντηση με ένα μειωμένο αριθμό χωρών εταίρων. Γιατί, γιατί η Γαλλία, η Ιταλία, η Γερμανία και η Ισπανία είναι οι χώρες που αυτή τη στιγμή έχουν αναλάβει δράση στην περιοχή του Σαχέλ. Και στην ασφάλεια και στην ενίσχυση αυτής και στην ανάπτυξη. Άρα λοιπόν ήταν ε, περιορισμένη σύνθεση στους κομβικούς παίκτες και που αυτή τη στιγμή ε, έχουν αναλάβει δράση στις χώρες του Σαχέλ. Είναι ξεκάθαρο, το είπε ο κύριος Μακρόν, πως είναι στο πλαίσιο της συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει κινήσει τη διαδικασία αυτή και γι' αυτό είχαμε την παρουσία της κυρίας Μογκερίνη και η οποία ήταν πολύ σημαντική. Νομίζω πως μίλησα για τα θέματα τα μεταναστευτικά. Θα ήθελα να μιλήσω τώρα για τα θέματα της εκπαίδευσης. και για τα όσα είπατε για ε, την ακτή του ελεφαντοστού. Λοιπόν, ναι, είναι πολύ δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο. Δεν μπορώ να μπω σε κάθε ε, παρουσίαση και να πω δύο λόγια για το κάθε project. Όμως, Έχουμε κάνει πολύ μεγάλες προσπάθειες για να ε, το βελτιώσουμε και αυτό τεκμηριώνεται. Ξεκινάμε με επιμόρφωση πριν τρέξει ένα project και πρέπει να σας πω πως έχουμε αυτές τις ερευνητικές δράσεις που μας επιτρέπει να προετοιμάσουμε όλα τα έγγραφα, να προετοιμάσουμε τη στρατηγική μας και την εκτέλεση για τη χρηματοδότηση των project και πρέπει να σας πω πως οι τόποι ε, που είναι προσπελα... Ε, τα, τα site που έχουμε ε, δίνουν ενημερωμένες πληροφορίες για το πώς τρέχει η εκτέλεση κάθε διαφορετικού project. Ξέρω πως χρειάζεται να κάνετε μια πιο σε βάθος ε, αναζήτηση. Είναι μόνο ένα εργαλείο η έκθεση η αιτήση αλλά έχουμε αυτό το site και ένα ακόμα site που θα ανοίξουμε σε μια εβδομάδα ή σε κάποιες εβδομάδες που θα σας δώσει λεπτομερείς πληροφορίες project ανά project για να μπορείτε να τα παρακολουθήσετε για μια φορά ακόμα να σας πω πως η ακτή του Ελεφαντοστού είναι μια χώρα, γιατί μιλήσατε για το Κοντιβουάρ, είναι μια χώρα καινούρια στο καταπίστευμα προς το παρόν κάνουμε αυτή τη στιγμή το διάλογο για τη μετανάστευση με τη χώρα αυτή και θα γίνει και μια ανάλυση για το ποια είναι η δράση η οποία θα είναι πιο στοχευμένοι για να τους χρηματοδοτήσουμε μέσω καταπιστεύματος. Μην ξεχνάτε πως αποτελεί μία απλή επιπλέον συνεισφορά σε σχέση με τα όσα κάνουμε για τις χώρες αυτές. Αν δείτε την ακτή του ελεφαντοστού θα δείτε πως έχουμε το εθνικό ενδεικτικό πρόγραμμα για τη χώρα αυτή και στο θέμα αυτό τονίζουμε την απασχόληση, τη δημιουργία απασχόλησης, τις επενδύσεις, τη διακυβέρνηση ε, και την βελτίωση της κυβέρνησης και του προπολογισμού της χώρας. Άρα λοιπόν θα τα δείτε και έχουμε και κάποια κονδύλια στο καταπίστευμα που θέλουν να δούνε ποιοι χώροι δεν καλύπτονται από το Εθνικό ε, Ενδεκτικό Πρόγραμμα και εδώ θα τα δείτε είναι ένα χώρα, έτσι ώστε να έχουμε κάτι το επιπρόσθετο σε σχέση με τους στόχους που έχουμε στο καταπίστευμα. Άρα λοιπόν, για την απασχόληση μπορούμε να έχουμε το εθνικό πρόγραμμα το οποίο ε, χρηματοδοτεί, άρα δεν το κάνουμε μέσω καταπιστέματος. Αν αντίθετα έχουμε ένα project το οποίο ε, θα ασχοληθεί με ζώνες, οι οποίες είναι ζώνες ε, προέλευσης μεταναστών, τότε εκεί ε, νομίζω ότι η προστιθέμενη αξία είναι η χρηματοδότηση από το καταπιστεύμα. Άρα λοιπόν στην αναλυτική, στη φάση ανάλυση χρηματοδότηση λαμβάνουμε υπόψη τι μπορούμε να κάνουμε στη χώρα μέσω του Εθνικού Ενδεικτικού Προγράμματος ε, του κανονικού ή του περιφερειακού ενδεικτικού προγράμματος και εντοπίζουμε τι μπορούμε να κάνουμε μέσω καταπιστεύματος γιατί είναι κάποιες δράσεις οι οποίες δεν εμπίπτουν στους στόχους που έχουμε στα ενδεικτικά προγράμματα ή γιατί είναι πολύ συγκεκριμένες οι ανάγκες χρηματοδότησης. Εδώ έχουμε τις ε, πληροφορίες Και στο Τσάντ όταν πάτε θα πρέπει να συνεργαστείτε με την αντιπροσωπεία μας εκεί που έχει τις πληροφορίες και που αναλύει τις πληροφορίες αυτές. Και θα σας δώσουν ό,τι στοιχεία θέλετε και για το project και για τους εταίρους μας. Τώρα για τις ΜΚΟ δεν έχω εδώ την κατανομή, αλλά η χρηματοδότηση σε μεγάλο βαθμό δίνεται σε ΜΚΟ που είναι διεθνής, αλλά που συνεργάζονται με τοπικές μη κυβερνητικές οργανώσεις. Και στην έκθεση θα σας έλεγα πως ο κατάλογος αναγράφεται, θα δείτε όλα τα project που έχουν εγκριθεί με την υπηρεσία ή τη ΜΚΟ που είναι υποχρεωμένη ε, να εκτελέσει αυτό το project, να θέσει σε εφαρμογή αυτό το project. Νομίζω ότι οι πληροφορίες αυτές είναι διαθέσιμες. Και το ίδιο θα βρείτε στο site μας. Ετήσει πληροφορίες, αλλά πληροφορίες οι οποίες ενημερώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα και που επαναλαμβάνω μπορείτε να βρείτε στο site. Για την τελευταία ερώτηση, για το πώς γίνεται η διαχείριση του Ταμείου, να σας υπενθυμίσω πως δεν αναφέρθηκα στο θέμα αυτό, γιατί το έχουμε παρουσιάσει τον Ιανουάριο, αλλά να σας πω πως για το καταπίστευμα έχουμε Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από κράτη-μέλη, δωρητές, που συνεισφέρουν στο καταπίστευμα, αλλά εκπροσώπους και των κρατών μελών κρατών μελών από την Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν συνεισφέρουν μεν, αλλά είναι ως παρατηρητές στο Διοικητικό Συμβούλιο. Και υπάρχει ε, υπάρχει επίσης εκπροσώπηση των χωρών εταίρων που επίσης ως νομικό καθεστώς έχουν το καθεστώς του παρατηρητή αλλά βρίσκονται στο Διοικητικό Συμβούλιο και στο Διοικητικό Συμβούλιο ε, πάντα καλούμε το Κοινοβούλιο και διεθνείς οργανώσεις που μπορεί να λάβουν κάποιο κομβικό ρόλο για την συζήτηση συγκεκριμένων θεμάτων. Εκτός λοιπόν από αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο έχουμε επιχειρησιακές επιτροπές συγκεκριμένες για κάθε θηρίδα. Και εκεί έχουμε τα κράτη-μέλη που συνεισφέρουν και των ε, χωρών ε, που λαμβάνουν τη χρηματοδότηση. Και πρέπει να σας πω πως πολλές φορές κάποια ανάλυση που γίνεται μας οθεί στο να προκρίνουμε μία πρωτοβουλία. Κοιτάμε δηλαδή τα project τα οποία χρηματοδοτούνται, κοιτάμε τον Ήγηρα, τι χρηματοδοτούμε στο Αγκαντές και δεν περιμένουμε απλώς να έρθουν κάποια καλά project από μία καπάω μικρόν. Πολλές φορές δημιουργούμε εμείς, αν θα την πρωτοβουλία, γνωρίζοντας ποιες και εντοπίζοντας ποιες είναι οι ανάγκες γιατί εντοπίζουμε τις ανάγκες και απευθύνουμε μια έκκληση ή σε καπαόμικρον ή σε φορείς να μας προετοιμάσουν τα συγκεκριμένα project. Άρα λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν διαχειρίζεται η ίδια τα project, γιατί εμείς χρησιμοποιούμε τους εταίρους τους που εφαρμόζουν και που, και που εκτελούν αυτά τα project και εμείς κατευθύνουμε, εγκρίνουμε, παρακολουθούμε ε, έτσι ώστε όλα να πάνε σωστά. Μιλήσατε για τα ΣΔΙΤ. Δεν θα πρέπει εκτός από αυτή την ε, εταιρική σχέση δημοσίου ε, και ιδιωτικού κόσμου να χρησιμοποιήσουμε και άλλα εργαλεία που έχει στη διάθεση της Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε τη νέα πρωτοβουλία με το επενδυτικό ταμείο ε, για την ανάπτυξη και θέλουμε να προωθήσουμε όλες τις ιδιωτικές και δημόσιες πρωτοβουλίες οι οποίες από εκεί μπορούν να χρηματοδοτηθούν ε, είτε από αυτό είτε από κάποιο άλλο εργαλείο. Γι' αυτό δεν θα πρέπει να παριστάνουμε πως μπορεί τούτο το καταπίστευμα να τα καλύψει όλα. Πολλές φορές έχουμε επενδυτικά σχέδια τα οποία χρηματοδοτούνται από άλλα εργαλεία χρηματοπιστωτικά με τις νέες αυτές πρωτοβουλίες, με το ε, Ταμείο ανάπτυξη και με άλλες πόρους που έχουμε διαθέσιμους. Ελπίζω για τον πρώτο γύρο ε, απαντήσεων να σας έχω καλύψει. Άλλοι έξι. Λέει η Πρόεδρος, έχουμε άλλα έξι άτομα που έχουν ζητήσει το λόγο. Επόμενοι ομιλητέ. Ο κύριος Ρούμπιχ. Και μετά τον Πόλ ε, θα έχουμε την κυρία Λίτ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και νομίζω ότι η παρουσίαση αυτή είναι πάρα πολύ ωφέλιμη για όλους μας, γιατί έτσι βλέπουμε πώς στην πράξη de facto εφαρμόζονται τα πράγματα αυτά. Έχω δύο ερωτήσει να κάνω. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχαμε ξεκινήσει δύο προπαρασκευαστικές δράσεις. Η μία δράση είναι η επιχειρηματικότητα των μεταναστών, πώς μπορούμε δηλαδή να προωθήσουμε και να καθιερώσουμε την επιχειρηματικότητα στους μετανάστες και σε ό,τι αφορά την συνεργασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην ε, Αφρική με μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Ευρώπης. Θεωρώ ότι πρόκειται για ένα σημείο εστίασης στο μέλλον, το οποίο έχει πολλά να προσφέρει. Δεύτερο θέμα είναι η επιχειρηματικότητα των γυναικών. Πώς μπορούμε να προωθήσουμε τις γυναίκες, τις μητέρες και να τις ε, κάνουμε να προσεγγίσουν αυτή την οτροπία της επιχειρηματικότητας προκειμένου και αυτές να δραστηριοποιηθούν και να μην περιορίζονται στα οικογενειακά τους κατοίκοντα, να ξεπερνάνε και να συμμετέχουν στην οικονομική ζωή πραγματικά. Ο δεύτερος μεγάλος τομέας που με ενδιαφέρει είναι κατά πόσον υπάρχει κάποια στοιχεία τα οποία να μας επιτρέπουν να δούμε τι επενδύονται στις υποδομίες σε ό,τι αφορά την ίδρυυση, τις αποχετεύσεις, ε, τη σχετική τεχνολογία και για την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Υπάρχει λοιπόν κάποια παρουσίαση των στοιχείων για να δούμε τι πηγαίνει πού και τι μπορούμε να κάνουμε τα επόμενα χρόνια, τι προγραμματίζεται να γίνει τα επόμενα χρόνια. Σας ευχαριστώ ο κύριος Λίτς και μετά ε, η κυρία αλλά Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ θα μιλήσω γερμανικά. Η παρουσία σήμερα το πρωί νομίζω ότι μας κατέδειξε εκ νέου ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ περίπλοκη και δύσκολη, σαν να έχουμε δημιουργήσει ένα παράλληλο κόσμο. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω πώς όλα αυτά εντάσσονται στις γενικότερες ευρωπαϊκές δραστηριότητε μας. Το παράδειγμα, για παράδειγμα, του Παρισιού. Πολύ ενδιαφέρον ότι συμπεριλαμβάνονται υπηρεσίες που μπορούν και σε άποψη περιεχομένου να συνεισφέρουν το μάθαμε και από τον τύπο. Εμεί ω ε, βουλευτέ το μάθαμε από τον τύπο το τι συζητήθηκε στην Παρίσι. Νομίζω ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη να είναι σε ένα σύνολο και να μην υπάρχει μια παράλληλη δομή. Γιατί νομίζω ότι στη τελική ανάλυση και οι πόροι είναι πολύ περιορισμένοι. Χρειάζονται 20-30 ε, δισεκατομμύρια προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα θεσμηματα αυτά. Αλλά σε ό,τι αφορά τα θέματα εκπαίδευσης και κατάρτισης αναρωτιέμαι τι γίνεται σε ό,τι αφορά και τον κλάδο, το, τη διάσταση της ε, βιωσιμότητας. Ε, πού υπάρχει αυτή η σύνδεση με την Ευρωπαϊκή Αναπτυξιακή Βοήθεια. Πού απέτυχαν ε, τα κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, την συγχρηματοδότηση. Θα πρέπει να υπάρχει, λοιπόν, συνεκτική συνεργασία και με τις ΜΚΟ, αυτό που προσπάθησαμε να κάνουμε και στο Παρίσι. Μία ερώτηση. Ένα σημαντικό θέμα στο οποίο δεν αναφερθήκατε. Στις στρατηγικούς σας προσανατολισμούς ε, βασίζεστε και προσανατολίζεστε σε ό,τι αφορά και τους ε, βιώσιμους αναπτυξιακούς στόχους, όπως έχουν τεθεί. Για να μιλήσουμε και για το ευρύτερο πλαίσιο συνεργάζεστε με την ΕΑΖΟ. Πήγαμε και στη Μάλτα. Είδαμε τι γίνεται και με τις χώρες ΑΚΕ. Υπάρχει και εδώ μεγάλη παραπληροφόρηση. Πώς ε, συνεργάζεστε με την ΕΑΖΟ. Υπάρχει συνεκτική συνεργασία. Τελευταία ερώτηση. Τι γίνεται, για παράδειγμα, είπατε ότι οι κρατικές ε, οργανώσεις υποστηρίζονται. Τι γίνεται όμως με τα θέματα καλής διακυβέρνησης. Και για να αναφερθώ σε αυτό που είπε η κυρία Μακέβεν. Χρειαζόμαστε... Χρειαζόμαστε συναπόφαση του Κοινοβουλίου, πράγματι. Και γι' αυτό λοιπόν και από δική μου πλευρά ε, απευθύνω μεγάλη έκκληση να επιτρέψετε στους ε, βουλευτές να συμμετέχουν και να δημιουργούνται ε, δομές ε, οι οποίες να λειτουργούν στην εβδομάδα και όχι το Σαββατοκύριακο προκειμένου να μπορούμε να συμμετέχουμε κι εμείς. Μάλιστα λέει η Πρόεδρος. Η κυρία Χάουταλα. Να σας πω ποιο είναι στο κατάλογο. Um, next is Heide Hautala, and then it'll be Doru αυτοί λοιπόν είναι που έχουν το λόγο γιατί θα κλείσω τη λίστα γιατί δεν έχουμε και χρόνο συνάδελφοι. Πολλοί συναδελφοί ενδιαφέρονται για το θέμα αυτό και ενδεχομένω θα χρειαστεί να αφαιρέσουμε και κάτι από την ατζέντα. Να το μεταθέσουμε δηλαδή σε μελετική συνεδρίαση. Η κυρία Χάουτελα. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Αν αυτή η ανταλλαγή απόφαση υποτίθεται ότι αποτελεί τμήμα του σημαντικού κοινοβουλευτικού ελέγχου για το καταπίστευμα για την Αφρική, εγώ πρέπει να πω ότι με πιο πολλές ερωτήσεις και ερωτηματικά φεύγω παρά ήρθα. Γιατί ο έλεγχος δεν έχει να κάνει με αναφορά και παραπομπή σε κάποια ιστοσελίδα και σε στοιχεία αριθμητικά. Εγώ θέλω να ξέρω συγκεκριμένα, για παράδειγμα, οι θέσει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από το ψήφισμα του 2016 πώς έχουν ληφθεί υπόψη και πώς έχουν εφαρμοστεί σε ό,τι αφορά την, ε, το σχεδιασμό, την παρακολούθηση των προγραμμάτων. Να αναφερθώ σε μερικέ δηλώσεις για να έχουμε μια ιδέα το τι ήθελε και το τι ήθελε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό, το Αφρικανικό καταπίστευμα. Θέλαμε να συμβάλλει στην υποστήριξη, στην προστασία των ευάλωτων μεταναστών και θυμάτων διακίνησης με ιδιαίτερη επικέντρωση στις γυναίκες και τα παιδιά. Πώς το πετύχαμε λοιπόν αυτό, το πετύχαμε. Επίσης στο ψήφισμα αναφέραμε ότι τα έργα που καλύπτονται από το καταπίστευμα δεν θα πρέπει να έχουν σκοπό την αγνόηση, αν θέλετε, των παραγόντων που σπρώχνουν τον κόσμο να μετακινηθεί. Θα πρέπει να δούμε και ποιος είναι αντικτύπος στα ανθρώπινα δικαιώματα και να δούμε τι γίνεται και σε χώρες με συστηματική παραβίαση των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Θέλαμε λοιπόν- θέλω λοιπόν να μας πείτε κατά πόσο αυτό πραγματικά τηρήθηκε στον σχεδιασμό και στην εφαρμογή των προγραμμάτων και πώς λαμβάνεται υπόψη τις απαιτήσει των κριτηρίων του ODA. Πέτυχε λοιπόν αυτό. Σας ευχαριστώ κύριε Σπρεντζούλικα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα αυτό. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν την κυρία Μοντέζη και ίσως να χρειαστούμε ένα κανόνα να μιλάει κάθε ένας μας μόνο δύο λεπτά γιατί κατά τα άλλα ε, φαίνεται ότι παίρνει πολύ χρόνο και το θέμα είναι πολύ σημαντικό. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω, τα έγγραφα αυτά διατίθενται, στη, μάλλον τα, τα οποία έχει η Επιτροπή για το καταπίστευμα, θα μπορούσαν να μας χορηγηθούν, γιατί είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει πραγματικός έλεγχος στις δραστηριότητες ε, του καταπιστεύματος. Θα πρέπει να υπάρχει πραγματικός έλεγχος και επί της Επιτροπής αυτής. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω κατά δεύτερον, να απαντήστε μας με σαφήνεια παρακαλώ. Βάσει ποιας ανάλυσης προκύπτουν και επιλέγονται όλα αυτά τα έργα. Και πώς υποστηρίζονται αυτές οι αποφάσεις και πώς εξασφαλίζουμε ότι γίνεται σεβαστή σχετική νομοθεσία. Σας ευχαριστώ και σας ήταν πάρα πολύ συνοπτικό στις ερωτήσεις σας. Σλάιν, και Ευχαριστώ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Μοντέζη, την δόκτωρα Μοντέζη, για την παρουσίασή της που ήταν τόσο πλήρης. Όμως πρέπει να πούμε ότι η άποψη του ελέγχου που μπορεί να ασκήσει το Κοινοβούλιο είναι τελείως ανεπαρκής και οι εκθέσεις, οι αιτήσει και οι μηνύες δεν δίνουν αρκετές πληροφορίες για να αξιολογήσουμε τα επιμέρους προγράμματα και την συμβατότητά τους με, την, ε, με τις προτεραιότητες της ανάπτυξης, την καταπολέμηση της φτώχειας και τα κριτήρια και τους κανόνες του Ταμείου για την στήριξη καταπολέμηση θελωτμάτων ανάπτυξης δίκαιο έχει συνάδελφος Αρχεντίνη. Γιατί δεν περνάει ε, η δράση από τις παρουσιακούς οδούς ε, και γιατί ε, δεν συνδυάζονται οι δράσεις όπως παλιότερα. Αυτό που να δικαιολογήσει το διαπίστευμα Παίρνουμε κονδύλια που απευθύνονται, ε, έχουν ε, στόχο την ανάπτυξη και η Ευρωπαϊκή Ένωση, αντί να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην βιώσιμη ανάπτυξη, καλύπτει εσωτερικέ ανάγκε κάποιων επιμέρου κρατών ε, με τη δικαιολογία ότι καταπολεμούνται έτσι οι πηγέ τη μετανάστευση. Χρειάζεται λοιπόν τεκμηρίωση και συγκεκριμένη εκπόνηση εγγράφων από το καταπίστευμα. όπω είπε και ο συνάδελφο Φρουντζούλικα, γιατί δεν υπάρχουν δημόσιες συζητήσεις, γιατί δεν υπάρχει καμία συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών. Εδώ δεν έχουμε καμία ενημέρωση. Φαίνεται ότι οι εθνικοί φορείς που πολλές φορές βρίσκονται σε ανταγωνιστικές σχέσεις μεταξύ τους είναι αυτοί που ασχολούνται περισσότερο και αναλαμβάνουν την εκτέλεση των προγραμμάτων. Αυτό όμω πώς εξασφαλίζει την ανάληψη ευθύνη από τις ίδιες χώρες και επίσης για τους τοπικούς φορείς. Το 20% το αναλαμβάνουν με κυβερνητικέ οργανώσει. Φαντάζομαι μεγάλε παγκόσμιε με κυβερνητικέ οργανώσει. Οι τοπικοί φορεί, ποιοι είναι, ποιοι είναι αυτοί οι δικαιούχοι που τόπου αναλαμβάνουν τα προγράμματα. Και για την δουλειά τη ομάδα μα και τη επιτροπή μα. Επιμένουμε στη σωστή χρήση αυτών των κομπηλίων. Φαίνεται να υπάρχει απόλυτη έλλειψη ισορροπία τη εκπόνηση προγραμμάτων σε σχέση με τον στόχο καταπολέμηση τη λαθμετανάστευση ε, στα σύνορα και Φαίνεται, όπως ε, υπόθηκε στο ε, Παρίσι, τα σύνορά μας αντί να τα προστατεύουμε εδώ, τα πηγαίνουμε και τα μεταθέτουμε όλο ένα και νοτιότερα, στη Λιβύη, ε, στον Νίγηρα και στο Τσάντ. Εδώ λοιπόν η ταχύτητα των κονδυλίων του καταπιστεύματος φαίνεται να έχει εξυπηρετήσει την αιμονή των κρατών μελών με την ασφάλεια και την κατα την προστασία των εξωτερικών συνόρων. Για την περιφερειακή σας τώρα δράση υπάρχει σοβαρός αντικτύπος στις τοπικές οικονομίες. Και μας δώσετε το παράδειγμα του Νίγηρα. Σας ερωτώ το αν να χρηματοδοτούνται κέντρα πληροφόρησης που ε, χρηματοδοτούνται από την UM. Πώς πετυχαίνει να αποτρέψει τη μετανάστευση. Πώς εκριζώνεται η φτώχεια. Και πώς γίνεται να ε, επιτυγχάνονται αυτοί οι στόχοι χωρίς επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια ODA. Δεν παίρνουμε τους μετανάστες ε, και να τους στέλνουμε πίσω στα σπίτια τους. Δεν είναι καταπολέμηση της φτώχειας και των γενοσουργών αιτίων της λαδομετανάστευσης. Δηλαδή, Ευχαριστούμε κύριος Γκερέρο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα καταρχήν να με συγχωρέσετε που δεν ήμουν από την αρχή της ε, συνεδρίασης για την παρουσίαση και για το πρώτο τμήμα της συζήτησης. Συζήτησα το λόγο γιατί ήθελα να μιλήσω για το Παρίσι και τη διάσκεψη εκεί. Άκουσα κάποιες παρεμβάσεις οι οποίες αναφέρθηκαν στο θέμα αυτό και δεν είναι τόσο πολύ ερώτημα όσο πιο πολύ ένα αίσθημα ανησυχίας που με διακατέχει, γιατί κάποια από τα στοιχεία τα οποία συνδέονται με την ε, ε, συνάντηση στο Παρίσι γιατί θα πω πως αφενός είναι σημαντικό το ότι οι τέσσερις πιο μεγάλες οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, συναντιόνται και προσπαθούν από κοινού να βοηθήσουν και να δώσουν περισσότερες ευκαιρίες στην Αφρική και όλα αυτά, αλλά κάποια στοιχεία θα πρέπει να αναλυθούν και να μας ανησυχούν. Δηλαδή, εκτός από ε, τις συνεντεύξεις τύπου και τα ανακοινοθέντα, ε, νομίζω πως η στόχευση είναι περισσότερο η μετανάστευση και όχι η ανάπτυξη. Δηλαδή, νομίζω πως για μας και για την πλειοψηφία του Κοινοβουλίου, το επιβραδύνουμε την ε, λάθρο μετανάστευση δεν είναι στόχος αλλά αποτέλεσμα. Αποτέλεσμα μιας δράσης η οποία θα δώσει ευκαιρίες στις χώρες προέλευσης και στις χώρες διέλευσης. Αν δηλαδή δεν έχουμε ως στόχο να φρενάρουμε την ε, μετανάστευση, θα πρέπει να κάνουμε κάτι το οποίο θα φέρει θετικά αποτελέσματα, θα δώσει ευκαιρίες στις χώρες αυτές και νομίζω πως η Σύνοδος στο Παρίσι ασχολήθηκε περισσότερο με τη μετανάστευση, μια και οι περισσότερες χώρες που συμμετείχαν αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν μαζικές αφήξεις μεταναστών και προσφύγων. Το δεύτερο που με ανισχύει είναι η σύγχυση που δημιουργήθηκε. Δηλαδή, εάν έχουμε το εργαλείο με αυτά τα καταπιστεύματα. Γιατί να δημιουργήσουμε και άλλα παράλληλα συστήματα, άλλες παράλληλες εναλλακτικέ δράσεις. Τρίτον, στη χρηματοδότηση. Γιατί το καταπίστευμα, όντως, στο μεγαλύτερο βαθμό χρησιμοποιεί ευρωπαϊκά εργαλεία, φορές κρατών μελών, είναι ένα πολύ μικρό τμήμα, 200 εκατομμύρια ευρώ νομίζω είναι. Και όσο έχουμε project ε, ομαδικά χωρών και όχι όλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η χρηματοδότηση θα τίνει να εξαφανίζεται και να προκρίνονται περισσότερο πολυμερή ή διμερή ε, project, όχι όμως κοινοτικά. Και τέλος, αυτή η δράση περιορίζει τη δυνατότητα που έχει το Κοινοβούλιο να ελέγχει με ποιο τρόπο ε, εφαρμόζονται οι πολιτικές, οι αναπτυξιακές, γιατί εθνικοποιούνται. Και όταν δεν εθνικοποιούνται, νομίζω ε, αντιστοιχούν σε ομάδες κρατών μελών, πιο περιορισμένες. Θα πρέπει να παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις αυτές με όλες τις πρωτοβουλίες που τις βλέπουμε σε πολλούς χώρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, ομάδες χωρών και κρατών μελών με αποτέλεσμα να αποδυναμώνεται η συνολική σφαιρική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, ευχαριστούμε. έχω μια ερώτηση για τη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου και θέλω να καταλάβω σε τι βαθμό η αρχή της εταιρική σχέσης είναι αρχή που καθοδηγεί τη δράση του Διοικητικού Συμβουλίου το Διοικητικό Συμβούλιο έχει συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των κρατών δωρητών και των δικαιούχων κρατών που είναι εκεί ως παρατηρητές. Η ερώτηση μου λοιπόν είναι, ας πάρουμε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, μια δράση που στόχο έχει να γίνει κάτι στο Μάλι και πρέπει να λάβει απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γαλλία μπορεί να βρεθεί σε θέση ε, ε, μειοψηφία. Παρόλο που είναι μια χώρα που έλαβε δράση ε, στο Μάλι που σταμάτησε την τρομοκρατική δράση στα 50 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Μπάμακο που έκανε ό,τι μπορούσε. Τι θα συμβεί σε αυτή την περίπτωση, είναι παρανόηση, Ποιο είναι ο πραγματικό ρόλο των χωρών δικαιούχων. Λέτε ότι έχουν ρόλο παρατηρητών. Αλλά μιλάμε για εταιρική σχέση και οι δικαιούχοι θα έχουν την κουβεντούλα τους να πούνε. Είναι απλώς λοιπόν παρατηρητές από, στα θέματα που προβλέπει να συζητήσει το Διοικητικό Συμβούλιο ή συμβαίνει κάτι άλλο στην πράξη. Έχουν μήπως άλλη βαρύτητα οι δικαιούχοι στο πλαίσιο αυτό. Και τελευταίο ερώτημα. Σε ό,τι αφορά αυτό το καταπίστευμα που στο γενικότερο πλαίσιο της αναπτυξιακής ε, βοήθειας. Πώς γίνεται η σωστή επιλογή μεταξύ των δράσεων που μπορεί να είναι προσοδοφόρες, αλλά δεν ε, καταλήγουν άμεσα στην εξάλληψη της φτώχειας, σε σύγκριση με άλλα προγράμματα τα οποία ε, στοχεύουν απευθεία στην εκρίζωση της φτώχειας, αλλά δεν είναι ε, αναγκαστικά προσοδοφόρα. Διότι είναι δύσκολο να καταπολεμηθεί η φτώχεια. Σε μια αναπτυσσόμενη χώρα δεν μπορεί να αναπτυχθεί το ΑΕΧ χωρί να υπάρξει κανένα αντίκτυπο, καμία επίπτωση στην εκρίζωση τη φτώχεια. Πώ γίνεται λοιπόν η σωστή επιλογή. Ωραία. Πολλέ ακόμη ερωτήσει. Προσπαθήστε να είστε τηλεγραφικοί. Έχετε παρόμοιες ερωτήσει με τις προηγούμενες. Ε, πολλοί ρώτησαν περίπου το ίδιο. Εταιρική σχέση, λογοδοσία, συνάδελφοι. Με τα προβλήματα συνάντηση Διοικητικού Συμβουλίου της Παρασκευές έχουμε ανοιχτό διάλογο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ζητήσαμε να υπάρξει μετακίνηση των ημερομηνιών σε φάσεις που το Κοινοβούλιο συνεδριάζει, Δευτέρες πρωί, ε, όταν είμαστε στο Στρασβούργο, όλα αυτά έχουν ε, ληφθεί υπόψη. Κάποια ήδη επιλύονται, είναι πρακτικά. Κυρία Μοντές, ευχαριστώ. Για τις ερωτήσεις που αναφέρατε, Πρόεδρε, κάποιες φορές είναι πολύ ευρείες. Οπότε θα προσπαθήσω να είμαι κάπως συνοπτική για να μείνω εντό του χρόνου. Σε σχέση με τον ρόλο του Κοινοβουλίου. Είπα ξεκινώντα ότι είναι ξεκάθαρο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, φροντίζει στο έπακρο να υπάρξει ένα ξεκάθαρο ρόλο του Κοινοβουλίου. Ε, φροντίζει να υπάρχει επιπλέον πρόσβαση για τα μέλη του Κοινοβουλίου στις πληροφορίες για τους δικαιούχους των εθνικών λογαριασμών όπως έχουν εγκριθεί και για τους ετήσιους λογαριασμούς του ΦΕΔ. Φροντίζουμε όχι απλώς να γίνουν σεβαστά όσα γίνονται παραδοσιακά στα πλαίσια του ΦΕΔ, αλλά να εγγυηθούμε την σημαντική πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες είτε στη φάση την προπαρασκευαστική, είτε στην επόμενη. Δυστυχώ απουσιάσατε, τώρα το έδειξα στην αρχή και όλη τη διάρκεια τη παρουσίαση ε, που μπορείτε να έχετε, ότι υπάρχουν στοιχεία που διασφαλίζουν την διαφάνεια της πληροφόρησης για το Κοινοβούλιο. Υπήρξε και άλλη ερώτηση για την εταιρική σχέση στον κατάλογο των πιλωτικών προγραμμάτων έδειξα και ανέφερα τα πρώτα προγράμματα που ανέφεραν την Σενεγάλη. Συνολικά, όταν κοιτάζω την περιπλοκότητα των προγραμμάτων, ε, ξαναλέω ότι 25% των κονδυλίων πρώτο σκοπό είχαν την ε, πρωτοβουλία των οικονομικών ευκαιριών για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Στα προγράμματα αυτά, που αποτελούν μία από τις πτυχές, υπάρχει στήριξη και για την δημιουργία, για την ε, υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, είτε με την επαγγελματική κατάρτιση, είτε με την οικονομική στήριξη, με τον εντοπισμό ενός προγράμματος, ενός business plan, το οποίο χρηματοδοτείται για νέα επενδυτικά προγράμματα. Πρόκειται για μια συνεισφορά περιορισμένη, διότι η ίδια η φύση του καταπιστεύματος δεν έχει σκοπό όλη έμφαση να δοθεί εκεί. Θέλει να ευνοηθούν οι εταιρικέ σχέσει, να ευνοηθεί το επιχειρηματικό περιβάλλον, η πρόσβαση των γυναικών, η οικονομική δράση. Αυτά είναι ε, θέματα κλειδιά τη αναπτυξιακή μα πολιτική, όπου απαντεί το σύνολο των διεκτικών προγραμμάτων των κρατών μελών και των επιμέρους γεωγραφικών περιοχών. Τέλος πάντων το καταπίστευμα αυτό δεν έχει την φιλοδοξία να κάνει τα πάντα. Είναι ένα καταπίστευμα λιγότερο από 3 δισεκατομμύριο. Δεν μπορώ να το συγκρίνω με τα 7 δις, εάν μιλήσουμε μόνο, μιλήσουμε για τη φυρίδα Σαχέλ και Δυτική Αφρική. 7 δις, ε, στη χειρότερη περίπτωση, για να βοηθήσουμε τους ιδιώτες, την απασχόληση, τις επενδύσεις. Το καταπίστευμα αυτό δεν μπορεί να τα κάνει όλα. Το ίδιο και για την ε, μόρφωση και την παιδεία. Η παιδεία θα συνεχίσει να παραμένει προτεραιότητα, προτεραιότητα που αναφέρεται στα εθνικά ενδεικτικά ε, προγράμματα και τα ενδεικτικά γεωγραφικά προγράμματα. Εάν υπάρξουν λοιπόν τμήματα του καταπιστεύματος που αφορούν την παιδεία, στην Ουγκάντα, στη Σομαλία ή στην Ερυθρέα, εκεί συγκεκριμένα βοηθάμε τα παιδιά των εκτοπισμένων που έχουν εγκαταλείψει το σχολείο να πάνε πίσω στο σχολείο, να ξαναπιάσουν την σχολική αγωγή. Αλλά δεν μπορούμε να ε, στοχεύσουμε το εκπαιδευτικό σύστημα συνολικά ή τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης στην εκπαίδευση. Πρέπει να διευκολύνουμε το σκέλος των εκτοπισμένων, των επιστρεφών των ε, λαθρομεταναστών. Αυτή είναι η πληθυσμή στόχος. Εκεί πρέπει να απαντήσει το καταπίστευμα, σε ένα στόχο που είναι πιο ε, συγκεκριμένος. Δεν μπορούμε να καλύψουμε όλους τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Για άλλη μια φορά λοιπόν, στην επιλογή των προγραμμάτων πρέπει να κάνουμε και κάναμε τη σωστή διασύνδεση και για αυτό το καταπίστευμα το διαχειρίζονται τρεις ομάδες, τρεις διαχειριστικές επιτροπές, οι ίδιες που ασχολούνται με τα επιμέρους γεωγραφικά και εθνικά ενδεικτικά προγράμματα, για να φροντίσουν να υπάρξει ε, συνδυασμός στη συμπληρωματικότητα των δράσεων και να επιδιωχθούν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης ή πιο συγκεκριμένοι, πιο περιορισμένοι στόχοι που έχουν να κάνουν με το καταπίστευμα το ίδιο. Για την επιλογή λοιπόν των προγραμμάτων γίνεται με βάση τον εντοπισμό των αναγκών. Κάθε πρόγραμμα έρχεται έτοιμο με μια ανάλυση για το ποια είναι τα προβλήματα. που θα εντοπιστούν στην πράξη, εντοπισμός των αναγκών που βασίζονται σε άλλες μελέτες, σε άλλες ερευνές που με τη σειρά τους διευκολύνονται από την ερευνά μας, όμως η ανάλυση των αναγκών όπως παρουσιάζεται περιλαμβάνεται πλέον στα προγράμματα. Οι στόχοι για να θεωρηθούν πρέπει να περιλαμβάνονται στα προγράμματα και σας έδειξα προηγουμένως πώς με το σύστημα παρακολούθησης που έχει δημιουργηθεί και αυτό είναι δουλειά της Επιτροπής βεβαιωνόμαστε ότι οι στόχοι που αναφέρονται στα προγράμματα όντως επιτυγχάνονται. Όλα αυτά είναι μέρος της διαχείρισης ε, της βοήθειας. Τώρα, για το Παρίσι. Οι συζητήσεις στο Παρίσι επικεντρώνονταν σε ένα σημείο. Αλλά το θέμα είναι που βρισκόμαστε σήμερα. Σήμερα ε, θέλουμε να έχουμε πρόσβαση στη Λιβύη, στις ε, με παραμεθόριες περιοχές της Λιβύης. Σήμερα ο, ο ΙΕ και η Πατηρομοστία ανακαλύπτουν καταβλισμούς ε, εγκλεισμένων θα έλεγε κανείς προσφύγων. Δείτε οποιοδήποτε ρεπορτάζ ε, στα διεθνή μέσα και θα δείτε ότι η κατάσταση είναι αυτή. Σήμερα λοιπόν στη Λιβύη έχουμε έναν σημαντικό αριθμό ανθρώπων οι οποίοι είναι καταλημμένοι σε συνθήκες εξαθλίωσης και ε, σε καταστάσεις λοιμού δεν είναι λοιπόν ο στόχο να σταματήσουμε τη μετανάστευση στα σύνορα, είναι να αντιμετωπίσουμε ένα ανθρωπιστικό πρόβλημα, να δούμε πώ θα βοηθήσουμε όλα αυτά τα άτομα που βρισκόνται στι μεταναστευτικέ οδού. Αυτός, είναι και, είναι ο σκοπός της δράσης μας. με συγκεκριμένο στόχο πώς μπορούμε να παρέμβουμε και να αντιμετωπίσουμε τις περιπτώσεις ασύλου ε, άτομα που βρίσκονται σε συνθήκες εξαθλίωσης στη Λιβύη ή σε άλλα σημεία της μεταναστευτικής οδού προς την Ευρώπη. Βεβαίω υπάρχει μια διάσταση ασφάλειας, αλλά μην κρυβόμαστε από την πραγματικότητα. Είδαμε τι έγινε το καλοκαίρι στην Ισπανία, είδαμε τις τρομοκρατικές επιθέσεις και ξέρουμε σήμερα ότι υπάρχουν τρομοκρατικές δυνάμεις που εγκαθίστανται στις περιοχές του Σαχέλ, σε εγκαταλειμμένες περιοχές, εκεί που δεν υπάρχει καμία διακυβέρνηση. Το καταπίστευμα λοιπόν μεταξύ των στόχων του, ε, είναι σαφής ο στόχος αυτός, θέλει να παρέμβει και για τη σταθεροποίηση κάποιων περιοχών που είναι τελείως ε, εγκαταλειμμένες στο Σαχέλ. Ειδικά σε αυτό το τμήμα του Σαχέλ που είναι το σημείο διέλευσης από τις ε, χώρες νότια της Σαχάρας προς τη Βόρεια Αφρική και που εγκαθίστανται όλες εξετρομιστικές δυνάμεις και η διακίνηση και διακινητές από όπλα και ανθρώπους μέχρι ναρκωτικά και ό,τι άλλο θέλετε. Εδώ λοιπόν Πρέπει να ενισχύσουμε τις χώρες εταίρους για να αντιμετωπίσουν τις ίδιες ελλείψεις τους. Ελλείψεις στην ασφάλεια και όχι μόνο τους πόρους. Δεν υπάρχει λοιπόν αιμονή με την ασφάλεια, υπάρχει ένα στοιχείο, μια διάσταση ασφάλειας που είναι ένας κοινό στόχος των ε, χωρών εταίρων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορούμε αυτό να το απαρνηθούμε. Ε, τρίτο στοιχείο για το Διοικητικό Συμβούλιο και την εταιρική σχέση που αναφέρθηκε, πρέπει να σεβαστούμε και την νομιμότητα των όσων κάνουμε. Υπάρχει ένα οικονομικός κανονισμό ο οποίο μας καθοδηγεί. Ο οικονομικός κανονισμό απαιτεί στο Διοικητικό Συμβούλιο να συμμετέχουν επισήμως μόνο χώρες δωρητέ ω μέλη. Επειδή ακριβώ η ε, κατάσταση όμω είναι ε, εταιρική σχέση, περιλαμβάνονται και όλε οι χώρε εταίροι. Έχουν τον τίτλο παρατηρητέ, γιατί αυτό, που μας αυτό ακριβώ μα ζητά ο κανονισμό. Όμω, βεβαίω, εάν μπορούσατε να παρίσταστε στο Διοικητικό Συμβούλιο, θα βλέπετε ότι εργαζόμαστε με τι χώρε εταίρου σε ένα πλαίσιο πλήρου διαφάνεια και του δίνουμε για το λόγο. Οπότε, αν μια χώρα θέλει να συμβάλλει και να αναφέρει και πολύ συχνά το κάνει, γιατί είναι δραστήριε χώρε αυτέ, δεν είναι απλώς παρατηρητές ε, και τους φημώνουμε, μπορούν να παρέμβουν ε, και ενεργά στι συνόδου του Διοικητικού Συμβουλίου. Πρόκειται για ένα Διοικητικό Συμβούλιο που οι χώρε εταίροι έχουν ένα ρόλο παρατηρητού μεν, αλλά υπάρχει ε, ζωντανή εταιρική σχέση δε. Για την ώρα δεν χρειάστηκε να ψηφίσουμε ούτε σε Διοικητικό Συμβούλιο ούτε σε Επιχειρησιακή Επιτροπή, διότι αυτό που θέλουμε να πετύχουμε είναι να υπάρχει διάλογος και συνεισφορά ενεργός. Θετική συμβολή από το σύνολο των ε, δικαιούχων χωρών. Σας διαβεβαιώ ότι ως τώρα δεν υπήρχε καμία δυσαρέσκεια ούτε από κράτος μέλος ούτε από χώρα Είναι ανοιχτέ οι σύνοδοι του Διοικητικού Συμβουλίου και ελπίζω κάποια στιγμή το Κοινοβούλιο να μπορέσει να παρίσταται για να δει τι ε, σχέσει και τις ισορροπίες που διαμορφώνονται στο επίπεδο του Διοικητικού Συμβουλίου. Βεβαίως σημειώσαμε την ε, πρώτερη ενημέρωση ε, για τη συνόδους του Διοικητικού Συμβουλίου και ώστε το Κοινοβούλιο να μπορεί να πάρει μέρος, αν το θέλει, Δευτέρες και Παρασκευές για να διευκολύνουμε τη συμμετοχή σας. Και βεβαίως έχουμε και όλα τα έγγραφα τα οποία πρέπει να λάβουμε έτσι ώστε να κάνουμε έναν εκ των προτέρων έλεγχο και όχι απλώς να ενημερωνόμαστε. Δεν ξέρω, Σαρλ, θέλεις κάτι να απαντήσεις. Ξέρω πως έχουμε ε, χρησιμοποιήσει ήδη όλο μας το χρόνο και έχουμε καθυστερήσει, αλλά είναι σημαντικό το θέμα, οπότε ε, την έκθεση από τη Νέα Υόρκη θα την αφήσουμε για επόμενη συνεδρίαση γιατί θα πρέπει να συνεχίσουμε και την ε, ημερήσια ε, η ημερήσια διάταξη. Ήδη έχουμε καθυστερήσει μία ώρα για τους συναδέλφους από την ΕΚΟ ε, που περιμένουν να μας παρουσιάσουν τα δικά τους. Ε, για το θέμα που αναβάλλεται, εγώ γράφω την έκθεση, οπότε καταλαβαίνετε πως με αφορά περισσότερο, αλλά για τα θέματα της Νέας Υόρκης χρειαζόμαστε και εκεί χρόνο και είναι σημαντικό να δούμε και την έκθεση και τις προτάσεις και όλα τα σχετικά. Οπότε, το σημείο αυτό που είναι το σημείο 7 αναβάλλεται για μια επόμενη συνάντηση. Σάρλ, σας ευχαριστώ πολύ για την απάντηση που δώσατε για το πώς ε, ε, λειτουργεί και τη διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου. Βεβαίως και είναι συνενετικές οι αποφάσεις συνήθως, αλλά να δούμε τι θα γίνει σε περίπτωση συγκρουόμενων απόψεων. Πώς θα αποφασίσουμε, ποιος λαμβάνει την πρωτοβουλία του να αποσύρει μιας πρότασης. Ε, θα, πώς ψηφίζουμε, με πλειοψηφία, είναι ειδική πλειοψηφία. Τα κράτη-μέλη τα οποία είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ψηφίζουν ανάλογα με το βάρος και το μέγεθος της συνεισφοράς τους. Οπότε θα... Και τι γίνεται σε επίπεδο δικαιοδοσίας. Αυτά ήθελα να μου απαντήσετε. Η απάντηση είναι πολύ σύντομη. Έχουμε ε, τον εσωτερικό κατονισμό του καταπιστεύματος και όλα αυτά περιγράφονται. Οπότε, βεβαίω θέλουμε ένα συνενετικό πνεύμα, αλλά αν δεν μπορεί να βρεθεί, έχουμε τον πρόεδρο και τους κανόνες που επιτρέπουν να αποφασίσουν τον αριθμό ψήφων και επίσης το πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις. Οπότε δεν θα σας παρουσιάσω τώρα τη διαδικασία αυτή, ορίζεται με σαφήνεια στον εσωτερικό κανονισμό που δημιουργήθηκε με τη σύσταση του καταπιστεύματος, παρόλα αυτά ανεξάρτητα από τα δικαιώματα ψηφοφορίας και τα λοιπά, το πνεύμα που διέπει είναι αυτό της συνένεσης. Αν όμως υπάρξει πραγματικό πρόβλημα, όντως έχουμε κάθε δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε τα όσα υπάρχουν στον εσωτερικό κανονισμό και να γίνει με τον τρόπο αυτό η ψηφοφορία. Θέλετε κι εσείς, συνάδελφε, να πείτε κάτι. Ναι. Άρα λοιπόν είναι σημαντικό να έχουμε μία ε, εταιρεία διαχείρισης, μια επιχείρηση διαχείρισης που θα επιτρέπει να προετοιμάζονται τα project εν ώψη της απόφασης της Επιτροπής Επενδύσεων με το δικαίωμα να προτείνει ίδια και project, γιατί πολλά θα πρέπει να δημιουργηθούν από την αρχή. Υπάρχει, υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Οπότε στο site και στην έκθεση θα βρείτε την ε, περιγραφή του πώς λειτουργεί. Έχουμε το Διοικητικό Συμβούλιο έχουμε την Επιτροπή που λέγεται Επιχειρηστική Επιτροπή, αλλά είναι Διαχειριστική Επιτροπή και εκεί λαμβάνονται τα project και είναι υπεύθυνοι για κάθε θηρίδα έτσι ώστε γνωρίζουν ποια είναι τα δικαιώματα, ποιος, το έχει το δικαίωμα πρωτοβουλίας, ποιες είναι οι προτάσεις που έχουν υποβληθεί στην Επιτροπή αυτή προς χρηματοδότηση και η Επιτροπή αυτή, η διαχειριστική, κάνει και το monitoring και παρακολουθεί και τη συνέχεια κάθε τέτοια επιχείρησης. Άρα λοιπόν υπάρχει διαχειριστική επιτροπή. Αυτό που δεν υπάρχει είναι κάτι το οποίο επιτρέπει να ε, αναλαμβάνουμε δράση επιτόπου. Όχι, αυτό το κάνουμε μέσω εταίρων που μπορεί να είναι φορεί, μπορεί να είναι μη καπαόμικροι, που έχουν επιτόπου την ευθύνη. Η διαχειριστική αυτή επιτροπή, η επιχειρησιακή, έχει την διαχειριστική ευθύνη όλων αυτών. Πολύ ωραία. Έγινε πολύ καλή συζήτηση. Βλέπω πως οι συνάδελφοι, πολλοί συνάδελφοι, θέλουν να κάνουμε ερωτήσει για, για το Κοντιβουάρ, για παράδειγμα. μα έχετε κάνει πολλέ ερωτήσει. βλέπω την Έλλη, έχουμε τη νέα ομάδα εργασία για τη μετανάστευση. Ίσως θα μπορούσατε να πάρετε ένα-δύο παραδείγματα χώρα και να δείτε τι χρηματοδοτείται από το εθνικό ε, πρόγραμμα ε, το ανδεικτικό, τι δεν γίνεται, ποιε είναι οι συνέργειε, να μιλήσετε με κάποιου συναδέλφου και να μα δώσετε κανένα δύο παραδείγματα που μπορεί να αποδείξουν για ποιο λόγο εκκρεμούν κάποια θέματα. Και ποια είναι τα ευρύτερα θέματα που προκύπτουν. Γιατί είναι δύσκολο να τα δει κανεί απομονωμένα. Όπω είπατε και εσεί, είναι μικρό αυτό το χαρτοφυλάκιο σε σχέση με τα όσα κάνουν ε, γενικότερα για την περιοχή και νομίζω ότι για πολλέ χώρε είναι αρκετή η σύγχυση που προκαλείται από τα διαφορετικά ταμεία με τι διαφορετικέ ε, διατάξεις οπότε συνάδελφοι έγινε μια πολύ μεγάλη συζήτηση θα ευχαριστήσω την κυρία Μοντέση Προβλέπαμε 45 λεπτά, είναι δύο ώρες εδώ κοντά μας. Και με χαρά περιμένουμε να κάνουμε και κάποιες συναντήσεις όταν θα έχουμε τις ημερομηνίε έτσι ώστε να παρακολουθήσουμε τι γίνεται. Και σας παρακαλώ να μας τηρήσετε και ενήμερος. Σας ευχαριστούμε πολύ. So now, colleagues, we go back to item six. Περνάμε λοιπόν στο σημείο 6 της ημερήσιας διάταξης. Το 7, όπως σας είπα, θα το συζητήσουμε μια επόμενη φορά. Και τα 6, ε, σημεία 6 με 8 θα τα πούμε πριν το μεσημεριανό διάλειμμα. ανθρωπιστική κατάσταση στη Χέρα Λεόνη και στην Νοτιοανατολική Ασία. Συνάδελφοι από την ΕΚΟ, λυπάμαι που περιμένατε τόση ώρα. Ξέρετε όμως πως τα καταπιστεύματα και τα μεταφανιστικά είναι θέματα πολύ σημαντικά για μας, οπότε σας παρακαλώ πολύ να καθίσετε. Ήρθαμε τέλη Αυγούστου μετά τις διακοπές και βλέπουμε πως αντιμετωπίζουμε ανθρωπιστικές κρίσεις σε στιγμές που εμείς είχαμε την τύχη περισσότερο να είμαστε διακοπές και ακούσαμε όλοι τι συνέβη και στη Σιέρα Λεόνε. Σας παρακαλώ να μιλάτε πιο σιγά αν μιλάτε μεταξύ σας. Είχαμε ε, την, ε, όσα έγιναν στο Freetown του Σιέρα Λεόνε που επηρεάστηκε από τον έμπολα πριν από μερικά χρόνια και είχαμε τώρα κατολιστήσεις ε, και λάσπες που κατέστρεψαν την πόλη Έχουμε επίσης τον Νεπάλ, τη βορειοανατολική Ινδία, τον Μπαγκλαντές που επηρεάστηκαν από πλημμύρες 6 εκατομμύρια στον Μπαγκλαντές, 30 εκατομμύρια στη βορειοανατολική Ινδία και τον Νεπάλ. Άρα λοιπόν τεράστιες ανθρωπιστικές καταστροφές και θέλουμε να ξέρουμε πώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποκρίθηκε Έχουμε εδώ την κυρία Σμιτ που είναι από το γραφείο του ΟΗΕ για το συντονισμό των ανθρωπιστικών θεμάτων, η ΟΤΣΑ, από το γραφείο των Βρυξελών. Θα μας μιλήσετε εσείς για την απόκριση. Και έχουμε και τον κύριο Κραφ που είναι από τη Μονάδα για την Ασία, Λατινική Αμερική, Καραϊβική και ε, Ειρηνικό από την Γενική Διεύθυνση ΕΚΟ. Λυπάμαι ε, που καθυστερήσαμε, όμως θα καταπιστεύω ότι είναι σημαντικά και για τη δική σας δουλειά και ξέρω πως θέλετε κι εσείς να ακούσετε ε, τα όσα συμβαίνουν. Λοιπόν, δεν ξέρω ποιος θα ξεκινήσει. Κυρία Γκόλσμιτ φαντάζομαι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ ε, για που μου δώσατε το λόγο. Να σας πω πως θα ξεκινήσω ευχαριστώντας σας για τις δυνατότητες που έχουμε να, για να αντιμετωπίσουμε την πολύ δύσκολη κατάσταση πολλών ανθρώπων στο Μπαγκλατέ, στο Νεπάλ και στην βορειοανατολική Ινδία, όπως επίσης και τις κατολιστής της Σιέρα Λεόνε. Θα ξεκινήσω με την Ασία γιατί εκεί τα νούμερα είναι πραγματικά μεγαλύτερα. κατά τη διάρκεια των μουσώνων είχαμε τεράστιες πλημμύρες ε, και κατολιστήσεις. Μπαγκλαντές, Ινδία και Νεπάλ επηρεάστηκαν κυρίως. 41 εκατομμύρια άνθρωποι ε, πλήττονται στις χώρες αυτές. Άλλες χώρες στην Ασία επίσης επηρεάστηκαν, η Μιανμάρ, οι Φιλιππίνες και η Κίνα. Οι βαριές βροχοπτώσεις οδήγησαν σε απώλειες ανθρωπίνων ζώων, γύρω δηλαδή στους χίλιους θανάτους, τον εκτοπισμό ενός εκατομμυρίου ανθρώπων και την καταστροφή σχολείων, νοσοκομείων και ιδιωτικών οικειών. Σε πολλές περιοχές ακόμα δεν μπορούμε να φτάσουμε λόγω της καταστροφής των υπόδημων και παρόλο που η κατάσταση θα ε, ε, χειροτερεύσει επειδή συνεχίζονται οι βροχές, φαίνεται πως το όσο συνέβησαν στη διάρκεια των μουσώνων μπορεί να συγκριθεί με το τι γίνεται άλλες αντίστοιχες χρονιές. Ανησυχούμε ιδιαίτερα για τα θέματα υγείας. Εδώ αυξάνονται οι ανησυχίες δυστυχώς. Έχουμε πάρα πολλές μεταδοτικές ασθένειες που μεταδίδονται μέσω μόλυνσης των υδάτων και στο Μπαγκλαντές, τον Νεπάλ και την Ινδία ε, η, τα συστήματα ανταπόκρισης σε καταστροφές είναι πολύ ε, ε, έτοιμα να αντιμετωπίσουν ό,τι παρουσιάζεται, αλλά έχουμε και την προσφορά του Ερυθρού Σταυρού, της Ερυθρής η Μισελίνου, όπως επίσης και ιδιωτικών φορέων. Επίσης, να σας πω πως στην Ότσα έχουμε διορίσει ένα μέλος προσωπικού για να αντιμετωπίσει τα θέματα αυτά. Να σας πω πως στην Ινδία μέχρι τις 24 8 είχαμε 32,1 ε, εκατομμύρια ανθρώπους που επλήγησαν και 600 ε, άτομα περίπου έχουν τη ζωή τους. Μιλάμε για τις ε, πολιτείες Μπιχάρου, Ταρ και τα λοιπά στην στην Νοτιό στη βορειοανατολική Ινδία και να σας πω πως αυτή τη στιγμή έχει κινητοποιηθεί και ο στρατός για να βρει καταλήμματα. Η Ινδική κυβέρνηση είπε πως θα δώσει 312 εκατομμύρια δολάρια έτσι ώστε να προχωρήσουν σε δράσεις για ε, υποστηλώσεις ε, και για αποζημιώσεις. Ξέρετε πως ε, δέχτηκαν την προσφορά να στείλουμε και εθνικούς εμπειρογνώμονες για τεχνική υποστήριξη όσων περιοχών έχουν πληγεί από ε, αυτές τις πλημμύρες. 32 περιοχές στο ε, Μπαγκλαντές, στο βόρειο βορειοανατολικό και κεντρικό τομάτι, ε, κομμάτι επηρεάζονται πάνω από 8 εκατομμύρια άνθρωποι, 700.000 σπίτια σχεδόν καταστράφηκαν και 600.000 ε, άτομα περίπου βρίσκονται σε καταλήμματα έκτακτης ανάγκης. Από τι 27 Αυγούστου να σας πω πως έχουμε σημειώσει 40 θέματα και βεβαίω εκεί 40 θύματα και υπάρχουν προβλήματα ε, με το πόσιμο νερό, με τα τρόφιμα και με τις υπηρεσίες. Περιμένουν ακόμα ε, σημαντικές βροχοπτώσεις που θα δημιουργήσει περισσότερε πλημμύρε. Η κυβέρνηση του Μπαγκλαντέ έδωσε 820.000 δολάρια σε ξηρά τρόφιμα, σε ρύζι, σε σκηνές και σε χρήματα στις περιοχές αυτές. Ο, ο στρατός δεν έχει κληθεί, αλλά ε, χρειάστηκε να γίνει και μία ανάλυση ε, της κατάστασης από εμάς ε, μέσα Αυγούστου στις 10 κοινότητες που επηρεάστηκαν σε 10 περιοχές και τα ευρήματα χρησιμοποιούνται για τις συζήτηση που γίνονται μεταξύ διεθνών δωρητών και ανθρωπιστικών οργανώσεων. Έχαμε πολύ σημαντική πλημμύρα σε ε, που σημαντικής ε, πλημμύρες στο Νεπάλ με 1,7 εκατομμύρια ε, άτομα να επηρεάζουν. 460.000 άνθρωποι εκτοπίστηκαν και 19.000 άτομα αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε κάποιους άτυπους καταβλισμούς. Είναι οι 35 από 45 ε, περιοχές που ε, πλήγησαν και έδωσε βοήθεια ένα εκατομμύριο ε, ευρώ η κυβέρνηση του Νεπάλ έχει ζητήσει από την Ινδία βοήθεια 3,9 εκατομμύρια έχει πει πως θα διαθέσει η χώρα αυτή και ζήτησε και από άλλους διεθνείς δωρητές 25 Αυγούστου η δική μας ομάδα παρουσίασε ένα κοινό πρόγραμμα δράση με 49 εκατομμύρια ε, δολάρια προπολογισμό, ε, έτσι ώστε να προσφέρει ανθρωπιστική βοήθεια, καταλήματα, τρόφιμα, προστασία ζωή, εκπαίδευση ε, και ανάκαμψη για του επόμενου 6 μήνε. Η ομάδα μα αυτή τη στιγμή ήδη προετοιμάζει ένα σημείωμα για κάποιε δράσει διάσωση ανθρώπινη ζωή. Θα ήθελα τώρα να με επιτρέψετε να σα μιλήσω για τη Σιέρα Λεόνε όπου οι φοβερέ βροχέ δημιούργησαν κατολισθήσεις ε, έξω από τη Freetown τον Αύγουστο. Αυτό λοιπόν επηρέασε πάρα πολύ. 496 άτομα έχουν επιβεβαιωθεί ότι έχουν χάσει τη ζωή τους. Εκατοντάδες άτομα αγνοούνται και χιλιάδες έχουν μείνει χωρίς τα σπίτια τους. Και αυτό φυσικά έχει περιττέρω επιδεινωθεί από την, ε, τα προβλήματα χωροταξία και πολεοδομία και από την αποδάσωση, η οποία είναι ένα γεγονό. Και δυστυχώ υπάρχει διαρκή κίνδυνο για πλημμύρε, γιατί θα συνεχίσει η περίοδο των προπλογωτώσεων μέχρι τον Οκτώβριο. Και η Εθνική Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας έχει συντονίσει τις προσπάθειές της με υποστήριξη πολλών οργανώσεων του ΟΗΕ. WFPIA, WHN και με ΜΚΟ, με τον Ερθρό Σταυρό και με τους Ιατρούς Χωρίς Σύνορα και με την υποστήριξη του ιδιωτικού τομέα. Οι προσπάθειες έχουν επικεντρωθεί στην εντοπισμό των νεκρών και την παροχή πρώτων βοηθειών στους επιζησαντές. Υπάρχει αίτημα της κυβέρνηση του Σιελεόνε ναι, συγγνώμη, ζητώ συγγνώμη, ζητώ συγγνώμη η ομιλήτρια για την ταχύτητά τη. Υπήρξε λοιπόν έτοιμα από την κυβέρνηση της Χέρα Λεώνα για να μετά το έτοιμο αυτό αποστήλαμε και την ομάδα συντονισμού του ΟΗΕ που συναποτελείται από εμπειρογνώμονε διάφορων κρατών μελών η οποία και ε, σκοπό έχει να υποστηρίξει και την κυβέρνηση και τους συντονιστές σε ό,τι αφορά το συντονισμό των πληροφοριών και τις επικοινωνίες και το συντονισμό της βοήθειας. 5.900 άτομα ε, που βρίσκονται σε πέντε κοινότητες ε, και οι ανάγκες τους ε, εντοπίζονται σε ό,τι αφορά την ταφή των νεκρών, την παροχή τροφίμων, νερού, συστήματα υγειονομική περίθαλψης, παροχή τροφίμων και μη τροφίμων και άλλων ε, προϊόντων ε, στον κόσμο αυτό. Για παράδειγμα, να σας πούμε ότι έχουν δοθεί παροχή, έχει δοθεί τρόφιμα σε 2.500 νοικοκυριά. Η UNICEF επίσης ε, παρέχει ψυχοκοινωνική υποστήριξη και για τις μητέρες που θυλάζουν και στα παιδιά κάτω των 5 ετών σε ό,τι αφορά ή την BOE, την WFP, έχει αναπτυχθεί ένα εργαλείο από αυτές τις υπηρεσίες για την παρακολούθηση των αναγκών της κοινότητας ε, των πλημμυροπαθών. Υπό η UNICEF και άλλοι εταίροι παρέχουν ε, υποστηρίξη προς το Υπουργείο Υγείας, μεταξύ άλλων και ε, εκτίμηση των αναγκών, αλλά δεν υπάρχει Εντοπισμό κρουσμάτων χολέρας, αλλά η UNICEF ε, αναπτύξει, έχει αναπτύξει ένα σχέδιο για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων κρουσμάτων και επίσης ε, παρέχεται υποστήριξη προς το Υπουργείο και σε ό,τι αφορά την πρόληψη τέτοιων ε, λοιμόξεων. Ψυχοκοινωνική αρρωγή επίσης παρέχεται στο, στην Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας και είναι Χιλιάδες άτομα που λαμβάνουν τέτοια υποστήριξη και αρρωγή. Η άμεση ανταπόκριση στην καταστροφή αυτή ήταν ε, η απελευθέρωση ενός πακέτου 4,8 δισεκατομμυρίων εκατομμυρίων, συγγνώμη, για την επόμενη περίοδο των 10 μηνών. Στην παρούσα φάση οι ανάγκες φαίνεται ότι εστιάζονται πιο πολύ και στη μακροπρόθεσμη ανάκαμψη για να βρεθούν μόνιμες λύσεις ε, καταλήμματος για τους αστέγους, ε, μια εκτίμηση των ε, υγειονομικών αναγκών. Και στην παρούσα φάση υπάρχουν τέσσερα βασικά καταλήμματα. Προγραμματίζεται η κατασκευή δύο επιπλέον τέτοιων καταλήμματων, προκειμένου να υπάρξει ασφάλεια στην κατάλυση στα καταλήμματα αυτά η μετακίνηση των ατόμων αυτών στα καταλήμματα και στα νέα αυτά, στις νέες αυτές εγκαταστάσεις θα επιστρέψει και τη λειτουργία σχολείων σε ό,τι αφορά επίσης την παροχή χρημάτων, σε ό,τι αφορά την παροχή υπηρεσιών στα θύματα. Διάφορες οργανώσεις δωρητών έχουν οργανώσει α, παροχή βοήθειας προς την κυβέρνηση της Χεραλεών και πολλές εθνικές και διεθνείς οργανώσεις παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες το Ηνωμένο Βασίλειο 500 εκατομμύρια, η Ιρλανδία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Γερμανία, η Ισπανία, η οποία συνέβαλε με χρήματα αλλά και με μία ειδική ομάδα εμπειρογνωμόνων για τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση των θυμάτων. 8,3 εκατομμύρια δολάρια επιπλέον έχουν απελευθερωθεί από διάφορες οργανώσεις και χώρες για την παροχή υλικού εμπειρογνωμοσύνης επίσης σε διάφορους κλάδους. Και πρόεδρε, αγαπητοί βουλευτές, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας προσκαλέσατε και που αφιερώνετε χρόνο να συζητήσετε τέτοιες ε, κρίσεις οι οποίες ε, δυστυχώς δεν προσελκύουν την ε, διεθνή προσοχή αλλά κοστίζουν τη ζωή σε εκατομμύρια ανθρώπους. Θα δώσω το λόγο στον συνάδελφο για να μας μιλήσει για τα δικά του ζητήματα. Σας ευχαριστώ, ο κύριος Λάμπερτ λέει, η πρόεδρος. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους. Συνάδελφοι, αξιότιμοι βουλευτές, με χαρά βρίσκομαι εδώ σήμερα και θα ήθελα να συμπληρώσω τα όμως όμως είπε η συνάδελφος για την κατάσταση στην ε, Νότια Ασία σε ό,τι αφορά και την κατάσταση εκτακτού ανάγκης της Χεραλεόνη. Κυρία Πρόεδρε, είπατε ότι στις ε, είπα, μάλλον τα σχόλια που κάνετε για τις είπα ήταν πάρα πολύ επίκαιρα. Να επαναλάβω ότι υπάρχει μεγάλη προσοχή που αφιερώνεται στον τύπο για τα θέματα αυτά και βλέπουμε εδώ πέρα πλημμύρες οι οποίες επηρεάζουν περίπου 40 εκατομμύρια άτομα. Δεν είναι τσουνάμι, δεν είναι τεράστιος σεισμός, ούτε είναι ε, παγκόσμια κλίμακα καταστροφή φυσική. Αλλά πρόκειται για μια σημαντικότατη καταστροφή την οποία βλέπουμε να προβάλλεται πολύ περιορισμένα. Βλέπουμε ιδιαίτερα ότι αυτό ισχύει και για τις εικόνες στην τηλεόραση που φυσικά επηρεάζουν πάρα πολύ άμεσα και φυσικά η περιοχή την οποία συζητούμε είναι πιο δύσκολο να υπάρξει πρόσβαση σε αυτή, αλλά υπάρχει πρόσβαση. Αυτό ενδεχομένω να λέει και δύο λόγια για το ενδιαφέρον του κόσμου για τέτοιες καταστροφές οι οποίες λαμβάνουν χώρα σε περιοχές μακρινές, οι οποίες δεν αποτελούν επίκεντρο, αν θέλετε, της προσοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι στον ίδιο βαθμό όσο άλλες. Δεν υπάρχει αντίστοιχη κάλυψη από τη δημοσιότητα λοιπόν και από τον τύπο. Δεν θα ήθελα να επαναλάβω όλα τα σημαντικά στοιχεία τα οποία ακούσατε από την Ότσα. Έγιναν και κάποιες αποστολές επιτόπου προκειμένου να επαληθευτούν στο βαθμό του δυνατού φυσικά και η διεισόμαση τα στοιχεία αυτά και αυτά που μας αναφέρουν ε, διάφορες ε, οργανώσεις αλλά σε γενικέ γραμμέ πρέπει να ομολογήσουμε ότι τα αριθμητικά στοιχεία είναι ακριβή. Αυτά που μα παρουσίασε η ΟΤΣΑ, συμπεριλαμβανομένων και των ατόμων που βρίσκονται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκη. Να σα πω λοιπόν ποια ήταν η αντίδραση τη Γενική Διεύθυνση ΕΚΟ ω τώρα στην κρίση αυτή. Υπάρχει παρακολούθηση διαρκής του κέντρου παρακολούθησης της κρίσης, υπάρχει και παρακολούθηση επιτόπου στο Παγκλαντές και στην Ινδία. Έχουμε και μία μικρή κεραία, θέλετε, στο Νεπάλ. Τα παρακολουθούμε λοιπόν αυτά από την πρώτη ημέρα. Να αναφέρουμε ότι υπήρξε ταχύ αντίδραση στις ε, εκκλήσεις της Διεθνούς Νομοσπονδίας του Ερυθρού Σταυρού για να υπάρξει ε, κινητοποίηση του ντρεφ του ταμείου αυτού για την αντίδραση στις έκτακτες ανάγκες και Μιλάμε για 200.000 ευρώ, τις οποίες τα οποία και στην Ινδία στις ξηρασίες. Το ίδιο έγινε και το 2004 στο Νεπάλ. Είχαμε στείλει και πυρογνώμονες της ΕΚΟ επιτόπου στον Μπαγκλατές. Ολοκληρώθηκε η δικασία την προηγούμενη εβδομάδα στην Ινδία και στο Νεπάλ συνεχίζονται ακόμα οι εργασίες. Περιμένουμε αναφορά από τους συναδέλφους σήμερα και αύριο αντιστοίχω για να μας δώσουν την εκτίμησή τους. Και περιμένουμε φυσικά και την πλήρη τους έκθεση για την κατάσταση. Είχαμε επίσης ε, λάβει έκκληση της κυβέρνησης ε, του Νεπάλ για διεθνή αρρωγή και σε είδος αλλά και σε πόρους και η Απευθύνθηκε έκκληση στα κρατημέλη δεν υπήρξε αντίδραση από τα κρατημέλη για οποιαδήποτε τέτοια ανταπόκριση, για το οποίο είναι και κατανοητό, γιατί φυσικά υπάρχει και μεγάλο κόστος μεταφοράς σε ό,τι αφορά αυτά τα είδη πρώτης ανάγκης. Τρεις εκθέσεις ε, αντιμετώπισης κρίσεως έχουμε εκδώσει και οι βουλευτές έχουν, τα έχουν λάβει αυτά στο ESCC, τουλάχιστον αυτή είναι η συνήθιση διαδικασία σε περίπτωση κρίσεων. Η πρώτη αυτή έχει να κάνει θα δημοσιευτεί μάλλον στα τέλη της εβδομάδας με τα αποτελέσματα της ε, Επιτροπής Αξιολόγησης, τα οποία και θα ολοκληρωθούν. Με τα αποτελέσματα λοιπόν αυτά στο χέρι, θα εξετάσουμε ενδεχόμενο περαιτέρω υποστήριξη ε, στις χώρες αυτές που πλήττονται και στην περίπτωση του Μπαγκλαντές να σας πούμε ότι έχουμε ουσιαστικά δύο διαφορετικές ε, πλημμύρες. Η μία προς το Γάγκη, τον ποταμό Γάγκη, από τα σύνορα του Νεπάλ μέσα στο Νεπάλ, στα δυτικά του Μπαγκλαντές δηλαδή. Και στην δεύτερη περίπτωση έχουμε από τη Βόρεια Ινδία πλημμύρα, από το βορρά του Μπαγκλαντές. Και έτσι λοιπόν και οι δύο ποταμοί στο σημείο που συνενώνονται, οι πλημμύρες ήταν τόσο μεγάλες που τελικά κατέκλυσαν και πλημμύρισαν το 1 τρίτο της επικράτειας του Μπαγκλαντές. Μιλάμε για ένα 1,5 μέτρο νερού. Δεν ήταν τεράστιο το ύψο τη πλημμύρα, αλλά η έκταση τη πλημμύρα ήταν πραγματικά ανεπανάληπτη. Δεν το έχω ξαναδεί ποτέ. Ήταν τεράστια η έκταση που έχει πλημμυρίσει. Αυτό και πριν από τους μουσώνες. Αυτό μας ανησυχεί ιδιαίτερως, γιατί δεν έχει ακόμα τελειώσει η περίοδος των μουσώνων. Αυτό τι σημαίνει ότι θα πρέπει να περιμένουμε και περαιτέρω πλημμύρε και να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Αυτό που τονίζουμε είναι ότι ο... τα άτομα τα οποία έχουν πληχθεί στο Μπαγκλαντές και μιλάμε για πάρα πολλά άτομα, πάρα πολλά εκατομμύρια. Υπάρχει μεγάλη αντακτικότητα όμω από πλευρά του κόσμου. Είναι πάρα πολύ φτωχοί αλλά και αντακτικοί και έχουν συνηθίσει σε κάποιο βαθμό τι πλημμύρε. Είναι προετοιμασμένοι και θα πρέπει να το αναφέρουμε αυτό. Γιατί μετά από 20 χρόνια, χάρη στην ΕΚΟΝ, μετά από 20 χρόνια προγραμμάτων μείωση του κινδύνου σε περίπτωση κρίση, τελικά ο κόσμος θεωρούμε ότι είναι κάπως προετοιμασμένος. Έχουν, για παράδειγμα, τα έγγραφά τους, τις πράξεις τους, ε, τις πράξεις ιδιοκτησίας των σπιτιών τους, ε, τις ταυτότητές τους, σε πλαστικά α, κοιτία τα οποία και μεταφέρουν. Και στα σχολεία, για παράδειγμα, διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν τυχή κατά των πλημμύρων, ε, προκειμένου να μην είναι τόσο έντονος ο κίνδυνος τα έγγραφα φυλάσσονται πάντα σε ψηλά ράφια, απλά μέτρα, τα οποία όμως έχουν τεράστιο αντικτύπο σε περίπτωση πλημμύρα τέτοιου τύπου. Άρα πολλά σπίτια καταστράφηκαν, προφανώς ε, τα καταλήμματα και ε, η διαμονή των ανθρώπων αυτών αποτελεί πρώτο ζήτημα και φυσικά και η πρόσβαση σε καθαρά νερό αποτελεί πάντα βασικό ζητήματα γιατί προφανώς ε, τα νερά της πλημμύρας ε, μολύνουν πηγάδια, πηγές, τα υπόγεια ύδατα. Και χρειάζονται φυσικά και ε, υπηρεσίες υγιεινής. Αυτό που μας απασχολεί πιο πολύ είναι ότι σε κάποιες ε, περιοχές ε, έχουν καταστραφεί και οι σοδιές. Η επόμενη περίοδος σοδιάς είναι Οκτώβριος-Νοέμβριος. Δεν υπάρχει μεγάλο χρονικό διάστημα για να γίνει εκ νέου φύτευση. Και άμα συνεχιστούν και οι βροχές όπως προβλέπετε, θα χαθεί και η επόμενη σοδιά. Αυτή είναι μια κατάσταση την οποία ελπίζουμε να αποφύγουμε, γιατί υπάρχει φυσικά και θέμα επιστικής ασφάλειας ε, στο Μπαγκλαντές. Αυτές είναι λοιπόν οι πιο άμεσες ανάγκες που αντιμετωπίζουμε σε ό,τι αφορά τα καταλήμματα και την υγεία και την ε, πρόσβαση σε καθαρό νερό. Και φυσικά είμαι στη διάθεσή σας να απαντήσω σε οποιαδήποτε ερώτηση και θα ήθελα να αναφέρω και το θέμα της Μια καταστροφή άλλων διαστάσεων. 6.000 άνθρωποι επλήγησαν και εδώ από το Κέντρο Συντονισμού και Κατεπηγόντων δεν είχαμε κάποιον απεσταλμένο εκεί, πήγε κάποιος από τη Δυτική Αφρική για να δει δύο όμως τι έχει συμβεί. Και με δορυφορικές εικόνες από το σύστημα του Κοπέρνικου που χρησιμοποιεί το χρησιμοποιεί ο ΙΕ Παρακολουθήσαμε την ε, περιοχή που έχει πληγεί. τη συγκρίναμε με την προηγούμενη περιοχή. Εμεί έχουμε προβλήψει 340 εκατομμύρια ευρώ από τα μικρής κλίμακας εργαλεία αντίδρασης και η, το συμπέρασμα από την αποστολή εκεί ήταν ότι οι ανάγκες καλύπτονται από τη συμβολή μας και τη συμβολή άλλων χωρών Οπότε δεν ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός προστασίας πολιτών που θα χρειαζόταν από τα κάτι μέλη για να προσφέρουν έγκαιρη βοήθεια, εάν υπήρχε ανάγκη. Αυτά η πολύ σύντομη παρουσίασή μου και με στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε για αυτή την ε, επισκόπηση. Δεν είχαμε τόσες πληροφορίες στα μέσα, γιατί Σιέρα Λεόνε ναι. Αλλά για τα δυτικά της Νότιας Ασίας όχι. Ο κύριος Γκερέρο και η κυρία Χάουταλα. Ευχαριστώ πολύ για όλες τις πληροφορίες που μας δώσατε και για τις δράσεις σας και για την απόκριση για τις φυσικές αυτές καταστροφές και κυρίως για τη δουλειά που κάνετε προσπαθώντας να βοηθήσετε τον κόσμο τον οποίο επηρεάζεται από τις φυσικές καταστροφές αυτές, οι οποίες μπορεί και να συνεχίσουν, γιατί όπως είπατε αυτή τη στιγμή είμαστε στην εποχή των ε, μουσώνων. Οπότε μπορεί κανείς να σκεφτεί πως ενδεχομένως θα συνεχίσουν οι βροχοπτώσεις τις επόμενες εβδομάδες. Εδώ μιλάμε για φυσικές καταστροφές και πολλές φορές στην Επιτροπή Ανάπτυξη μιλάμε για συγκρούσεις, ο λοιμός σε κάποιες περιοχές του πλανήτη. που δημιουργείται από ανθρώπινους παράγοντες, άλλες φορές που προκαλούνται από φυσικές καταστροφές. Όμως, ο τρόπος για να αντιμετωπίσουμε τις καταστροφές εξακολουθεί να είναι πάντα μια ανθρωπιστική διαχείριση μιας κρίσης. Και αυτό εξηγεί Γιατί με τέτοιες τεράστιες ποσότητες βροχής όπως αυτές που έπεσαν στο Τέξας τα αποτελέσματα σε απώλεια ανθρώπινης ζωής είναι πραγματικά λυπηρά αλλά παρόλα αυτά είναι πολύ ε, χαμηλότερα από, τα, από τις συνέπειες που είχαμε στη Σιέρα Λεόνη ή στην Νοτιοανατολική Ασία. Και αυτό μας οδηγεί σε εξής σκέψεις. Πρώτα απ' όλα πως προφανώς ε, αντιμετωπίζουμε ε, μια κλιματική αλλαγή που θα φέρει πολύ πιο πολλές καταστροφές, πιο έντονες φυσικές καταστροφές και θα πρέπει η απόκριση που θα δώσουμε να το λάβει αυτό υπόψη, γιατί γνωρίζουμε σίγουρα πως θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδους φυσικές καταστροφές στο μέλλον ακόμα συχνότερα. Και δεύτερον, ο τρόπος με τον οποίο δημιουργήθηκαν αυτές οι πλημμύρες, αυτοί οι χήμαροι αποδεικνύουν τι, τι επιπτώσεις έχουν αυτές οι άτυπες συγκεντρώσεις πληθυσμού, αυτοί οι οικισμοί οι οποίοι δεν μπορούν να αντέξουν πλημμύρες και βροχές και τους οποίους θα μπορούσαμε να έχουμε προλάβει εάν είχαμε στρατηγικές μείωσης κινδύνου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Κοινοβούλιο στα πλαίσια του ΣΕΝΤΑΙ του 2015 και μέσω της Παγκόσμιας Πλατφόρμας του Κανκών της ίδιας χρονιάς έχουν ε, ε, υπογράψει κάποιες ε, δηλώσεις και εγώ θα ήθελα να πω κάτι, το οποίο, κάτι στο οποίο αναφέρθηκε και αναφέρθηκαν και εκπρόσωποι της ΕΚΟ για την αντιμετώπιση και τη μείωση κινδύνου σε τοπικό και σε εθνικό επίπεδο. Πιστεύω πως τέτοιου είδου δράσεις τη Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσαν να εντετικοποιηθούν πρώτον γιατί δεν χρειάζονται πολλούς πόρους ούτε οικονομικούς ούτε υλικούς και δεύτερον επειδή θα μπορούσαν να είναι πάντα έτοιμοι και να μην χρειάζεται μια απόκριση επίγουσας ανάγκη σε κάποια καταστροφή. Και τρίτον, επειδή θα πρέπει να ευαισθητοποιήσουμε τις αρχές για το γεγονός πως οι φυσικές καταστροφές πολλές φορές προκαλούνται από φυσικά φαινόμενα, αλλά οι επιπτώσεις τους μπορούν να απαλληθούν σε μεγάλο βαθμό ε, με προηγούμενη δράση. Ευχαριστώ. Πολύ σωστά αυτά που έλεγε ο Γκερέρο. Θα βλέπουμε λένε και περισσότερες τέτοιες καταστροφές, την έλλειψη προετοιμασίας, και το πλαίσιο προετοιμασίας ανθεκτικότητας στι ε, στις έκτακτες ανάγκες. Πρέπει αυτή την οξύ ανάγκη να την, να την αντιμετωπίσουμε και να σκεφτούμε τι μπορεί να κάνει το Ευρωκοινοβούλιο για να δώσει μια όθηση σε όλα αυτά. Στην ανθρωπιστική πλευρά οι προσπάθειες σας είναι αξιοθαύμαστες, παρόλο που οι πόροι ποτέ δεν εξαρκούν και αυτό πρέπει να το προσέχουμε στον προπολογισμό μας. Θα το συζητήσουμε και το απόγευμα αλλά έχω μια ερώτηση συστηματικά, πάντα την ίδια. Από αυτές τις ανθρωπιστικές δράσεις, ποιοι λαμβάνουν, πόσο λαμβάνονται υπόψη μάλλον οι ανάγκες των, ε, των ανθρώπων με ειδικέ ανάγκες γυναικών και παιδιών, των ανθρώπων με κάποιες ιδιαίτερες αδυναμίες. Ναι, κάποιες παρατηρήσεις και από τη δική μου πλευρά για την ανθρωπιστική απόκριση Αναφέρατε νομίζω ότι ένα από τα βασικά προβλήματα στη Σιέρα Λεόνε είναι η αποψήλωση και ο κακός ε, αστικός σχεδιασμός. Όταν τα είδατε, ε, πόσο βλέπετε να συμβάλλουν οι αναπτυξιακές μας πολιτικές στην αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων. Κατά την αξιολόγησή σας, μιλήσαμε πολύ για την ένταξη της ε, ανθρωπιστικής αναπτυξιακής βοήθειας το να τα παρακολουθήσουμε σε αυτή την περιοχή και επειδή είχαμε πει τα ξαναδούμε και έχουμε επενδύσει πολύ στο σύστημα υγεία τη Χέρα Λεών ε, στην προηγούμενη κρίση με τον έμπολα. Είδαμε να δίδονται πολλά χρήματα σε νοσοκομεία, κλινικέ κέντρα. Είδαμε στην τηλεόραση να χτίζονται μικρά νοσοκομεία σε κάποιες χώρες της Δυτικής Αφρικής. Ε, τι έχει μείνει από όλα αυτά. Βοήθησαν πουθενά. Οι επενδύσει αυτέ που έγιναν για να αντιμετωπιστεί ο έμπολα άφησαν πίσω τους κάτι. Έχουν, ας πούμε, οι άνθρωποι στη Σιέρα Λεόνα καλή πρόσβαση στην ε, υγειονομική περίθαλψη όταν συμβαίνει τέτοια καταστροφή. Ε, δεν βλέπω άλλοι συνάδελφοι να ζητούν το λόγο, οπότε ίσως να απαντήσετε. Ναι. Ίσως να ξεκινήσω εγώ. Έχετε πολύ δίκιο. Και θα συμφωνήσετε όλοι πιστεύω ότι Τέτοιε καταστροφέ μάλλον θα τι βλέπουμε συχνότερα στο μέλλον. Οπότε είναι σαφέ ότι οι προσπάθειε που γίνονται για την καταπολέμηση του κινδύνου των καταστροφών και τη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση του, πρέπει να ενταθεί. Επίση αληθεύει ότι η ευθύνη είναι και ευθύνη των ε, ενδιαφερόμενων αυτών χωρών. Το λέω και από την οπτική γωνία των διεθνών διαπραγματευσεών και του πλαισίου Σεντάι. για την αναγνώριση κάποιων ευθυνών. Πρέπει να αναλάβουν ευθύνε οι κυβερνήσει ε, όταν χτυπά μια καταστροφή σε εθνικό επίπεδο. Κάποιε από τι κυβερνήσει ακόμη δεν είναι έτοιμε. Το είδαμε με τον περασμένο τυφώνα στην Αϊτή τον Οκτώβριο. Η κυβέρνηση ήθελε να λάβει πρωταγωνιστικό ρόλο, αλλά ε, δεν είχε τις δυνατότητες. Όμως από την πρώτη στιγμή ανέλαβε ευθύνη στην περίπτωση της Ινδίας, στην περίπτωση του Μπαγκλαντές και του Νεπάλ. Η κυβέρνηση όντω έχει αναλάβει τον πρωταγωνιστικό ρόλο για την ε, εξέφραση μιας απόκρισης. Εγώ έχω εργαστεί πολύ καιρό στην Αφρική και έχω δει περιπτώσει που οι κυβερνήσει να λένε έχουμε πρόβλημα, ανοίγουμε τα σκύλα μα να βοηθήσει η εθνική κοινότητα. Σε κάποιε χώρε το βλέπουμε αυτό. Εδώ, όταν μιλάμε για εθνικέ καταστροφέ όλο ιδιαίτερω και ακόμη περισσότερο στην Ασία και τη Λατινική Αμερική, όπου υπάρχουν οι κυβερνητικέ δυνατότητε, και ολένα και περισσότερο και υπάρχει και ανησυχία για την προετοιμασία και την δυνατότητα αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, τα πράγματα είναι καλύτερα. Στην Ινδία δεν είναι ίσως όλοι πολύ πειθαρχημένοι με τις τοπικές κυβερνήσεις Έχουμε κάποια θέματα και αν με ζητήσετε τη γνώμη μου θα σας πω ότι μπορεί να υπάρξει διάλογος με την Ινδία για το θέμα αυτό. Η Ινδία όμως θέλει ανθρωπιστική βοήθεια. Όταν πήγαμε αποστολή στην Ινδία σε περασμένη περίπτωση, μια αποστολή παρακολουθήσεις γιατί υπάρχουν κάποια προγράμματα που τρέχουν, και θα εξέπνεαν στην Ινδία, στην ε, πρεσβεία μας είπαν ότι η Ινδία δεν θέλει ανθρωπιστική βοήθεια γιατί θέλετε να πάτε στην Ινδία, τι θα κάνετε, τι ανθρωπιστικά να δώσετε. Η Ινδία προσφέρει ανθρωπιστική βοήθεια. Υπάρχει δηλαδή πολύ μεγάλη δυνατότητα διακυβέρνηση που πρέπει να ενισχυθεί βεβαίω περαιτέρω, αλλά αυτό που μου δίνει η ελπίδα είναι ότι υπάρχει ευαισθητοποίηση ε, ιδίως στο Μπαγκλαντές ή με τους κυκλώνες στις ακτές του Μπαγκλαντές πριν από 5-10 χρόνια έχαναν τη ζωή τους εκατοντάδες χιλιάδες. Τώρα με 4.000 είναι τίποτα, μια χοφτά άνθρωποι είναι. Ε, διότι Ξεκίνησε ένα σύστημα γραπτών μηνυμάτων SMS, το οποίο άρχισε να προειδοποιεί γύρω στους ανθρώπους στην περίπτωση των κυκλώνων, τώρα λειτουργήσε και στην περίπτωση των πλημμυρών. Πρέπει να διατηρήσουμε λοιπόν αμύωτα τι προσπάθειέ μα, αλλά να τι συνεχίσουμε κιόλα για να συνεργαζόμαστε με τι τοπικέ κυβερνήσει και να βελτιώσουν τι δυνατότητέ του και την ετοιμότητά του και την απόκρισή του. Βέρα, θε να προσθέσει τίποτα. Ευχαριστώ Μάρτιν και εγώ θα ήθελα επίσης ε, να υποστηρίξω απόλυτα τα όσα ακούσαμε για την προστιθέμενη αξία και την ανάγκη να υπάρξει πρόληψη και φυσικά αυτό γίνεται από πλευρά του ΟΗΕ με την υποστήριξη όλων των κυβερνήσεων και με την υποστήριξη τη ότσο και φυσικά και σε άλλες ε, υπηρεσίε. και βλέπουμε επίση και την αξία τη. Ε, χρηματοδότησης ΥΠΕΚΟ και στην ΟΤΣΑ τονίζουμε πόσο σημαντική είναι η συνέχιση της ε, χρηματοδότηση αυτή σε επίπεδο που θα μας επιστρέψουν γιατί πρόκειται για ε, χρήματα τα οποία δεν είναι τεράστια αν θέλετε ε, αξία, αλλά έχουν μεγάλο αντίκτυπο και οι συναδελφοί μου στην DGECO νομίζω ότι μπορούν να πιστοποιήσουν την αξία των προγραμμάτων αυτών. Να συζητήσουμε λοιπόν τα θέματα αυτά και την πιο πολύ χρηματοδότηση, αλλά κυρίως και την επικέντρωση στην πρόληψη από πλευρά τη ΕΚΟ. Αυτό κάνει μεγάλη διαφορά πραγματικά. Θα ήθελα επίσης να αναφέρω και αυτό που είπα στην παρουσίασή μου, ότι όλες οι κυβερνήσεις ε, και υπήρξε και συνεννόηση και υποστήριξη μεταξύ των κυβερνήσεων από πλευρά τη Ινδία. Για παράδειγμα, υπήρξε οικονομική αρρωγή προ του ε, γείτονε. Φυσικά αυτέ είναι οι χώρε που έχουν την πρώτη ευθύνη και θα πρέπει να υπάρξει υποστήριξη. Αυτό σημαίνει και σε άλλα τμήματα του κόσμου. Σε ό,τι αφορά τα ευάλωτα, ευαίσθητα σημεία, και αυτό νομίζω ότι έχει να κάνει και αντιπροσωπεύει όλη την κοινότητα για ανταπόκριση στις έκτακτε ανάγκες. Φυσικά η ιδιαίτερη προσοχή στα προβλήματα αυτά και σε ό,τι αφορά την ανάληψη δράσεων θα πρέπει να πούμε ότι όλοι οι φορείς ε, προσέχουν ιδιαίτερα στους πιο ευάλωτους, τους ηλικιωμένους, τα παιδιά, τις γυναίκες. Α, αυτοί λαμβάνονται υπόψη κυρίως. Και εξασφαλίζουμε ότι πραγματικά λαμβάνουν υποστηρίξη. Και ο τρόπος που σχεδιάζονται τα πρόγραμματα σήμερα από τον ΟΗΕ μέχρι τη ΣΜΚΙΟ. Και παντού πάντα εξασφαλίζεται ότι δίνεται ιδιαίτερη προσοχή σε αυτά τα άτομα, στι ε, ομάδε του πληθυσμού και σε τέτοια θέματα όπω είναι η αποδάσωση. Να δώσουμε το λόγο και στην ε, Echo. Γιατί φυσικά ως ΟΗΕ υπάρχει το UNDP. Και εκεί θα λάβουν χώρα προφανώς στις συζητήσει. Ναι, ζητώ συγγνώμη πρόεδρε, ξέχασα να αναφέρω το θέμα αυτό. Εν συντομία για την ΣΕΡΙΑ Λεόντε. Νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ η συνεργασία με τους συναδέλφους από την DigiDevco, το οποίο είναι σε κάποιες περιπτώσεις πιο απλό και σε κάποιες λιγότερο απλό. Αλλά υπάρχει ένα διαρκής διάλογος σε κάθε περίπτωση και σε όλες ε, τις χώρες ε, σε παγκόσμιο επίπεδο, γιατί φυσικά υπάρχουν πιέσεις και στους προϋπολογισμούς. Η ΕΚΟ στο παρελθόν έχει ε, λάβει αιτήματα να χρηματοδοτήσει ενέργειες που μπορούν να χρηματοδοτηθούν και από άλλα μέσα. Και σημαντικό είναι να υπάρχει πάντα μια συζήτηση προκειμένου να αφαιρεθούμε από την εμπειρία της ΕΚΟ σε τέτοια ζητήματα. Τώρα, σε ό,τι αφορά συγκεκριμένα το θέμα της αποδάσωσης, θα πρέπει να σας δώσω μια απάντηση στο μέλλον. Δεν έχω αυτή τη στιγμή μια συνολική επισκόπηση της κατάστασης. Μάλιστα, λέει η Πρόεδρος. Νομίζω ότι έτσι απαντήσαμε τις ερωτήσεις. Θα ακούσουμε την απάντηση για την αποδάσωση σε κάποια άλλη χρονική στιγμή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, λοιπόν. Και θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε και τους ανθρώπους που βρίσκονται εκεί επί τόπου, στους εμπειρογνώμονες και παρέχουν την βοήθεια. Είναι θετικό το γεγονό ότι αναφέρεται ότι οι κυβερνήσει των χωρών αυτών ε, σε πολλές περιπτώσεις είναι αυτές που παίρνουν τα ενία. Αυτό είναι σημαντικό. Θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία και συντονισμένη παροχή αρρωγή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για το ταξίδι που κάνατε μέχρι εδώ σήμερα. Σας ευχαριστούμε. Συνάδελφοι, να περάσουμε στο τελευταίο σημείο. Είχαμε συμφωνήσει ότι όσοι έχουν έρθει για το σημείο 7, την ενημέρωση από από την αποστολή της Νέας Υόρκης του υψηλού επίπεδου πολιτικό φόρουμ που το αναβάλουμε και μετά θα ε, έχουμε προτάσεις για το πώς θα παρακολουθήσουμε την υλοποίηση των ε, στόχων της χιλιετίας. Αυτά και τα δύο μας θα τα δούμε σε επόμενη συνεδρίαση για να προετοιμαστούμε και καλύτερα. Ε, τώρα είναι η στιγμή μετά τις καλύτερες διακοπές ε, και κάποιοι συνάδελφοι ζουν να μην ήταν και στην αίθουσα αυτή τη στιγμή. Τώρα περνάμε στο σημείο 8. Έτσι είναι η χρήση του ποινικού δικαίου για την καταπολέμηση του ξεπλήματος ε, μαύρου χρήματος και Ξέρετε πως αυτή τη στιγμή ετοιμάζουμε μια γνωμοδότηση για την ε, νομοθετική πράξη στην οποία ε, επικεφαλής επιτροπή, κύριε Επιτροπή είναι η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ όπου εκεί είχαμε τον ίδιο συνάδελφο που την έγραψε που κάνει και τη δική μας και καλό θα ήταν ε, αγαπητέ Ιγνάσιο να παρουσιάσει στους συναδέλφους τα όσα συμβαίνουν, εσύ τα καταλαβαίνεις καλύτερα και να μας πεις και ποια θέματα άπτονται της δικής μας ε, επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω Ιταλικά. Διότι εδώ επιστρέφουμε στους ε, καιρούς ε, τους φοιτητικού, τους δικούς μου, γιατί σπούδασα νομική και θα μιλήσω για θέματα δικαίου. Η βασική έκθεση λοιπόν, η έκθεση για την οποία είμαι υπεύθυνο και αρμόδιος στη ΛΥΜΠΕ έχει να κάνει περισσότερο με ποινικά θέματα, ε, νομοθετικά και είναι πολύ σημαντικό γιατί προσπαθεί να εναρμονίσει τα νομοθετικά συστήματα των κρατών μελών για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Τα συστήματα λοιπόν έρευνας και ανάκρισης των κρατών μελών, έτσι όπως είναι αποσυνδεδεμένα, επιτρέπουν την ελευθερία κυκλοφορία βρώμικου χρήματος και την ανταλλαγή του ώστε να χρηματοδοτούνται παράνομες δράσεις. Και στην ανταγωνιστικότητα και στο σύστημα το ποινικό, το εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, υπάρχει δυστυχώς αυτή η κακή νομοθέτηση να μην εντοπίζεται το πόθεν έσχες κάποιων κεφαλαίων και ο καθένα να μπορεί να έχει οικονομική δραστηριότητα. Πολλές, φορές, πολλές φορές όμως τα κεφάλαια αυτά που φτάνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εδώ επενδύονται στην άλλη αγορά είναι κεφάλαια παράν, παράγονται από παράνομες ε, πηγές σε αναπτυσσόμενες χώρες. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, παίρνει μεγαλύτερη σημασία και πρέπει να σκεφτούμε τι συμβαίνει στις αναπτυσσόμενες χώρες μέσω της οδηγίας, την έκθεση μάλλον της ΛΥΜΠΕ και αυτής που ετοιμάζουμε στην Επιτροπή Ανάπτυξης προσπαθούμε να βρούμε κάποιες λύσεις ώστε να διευκολύνουμε τους Ευρωπαίους δικαστές να έχουν τα εργαλεία στη μέση τους για να αντιμετωπίσουν, στην διάθεσή τους για να, για να αντιμετωπίσουν τα κεφάλαια που έρχονται από παράνομες πηγές. Διακίνηση ναρκωτικών, εμπορία ανθρώπων, διαφθορά και άλλου είδους παράνομες δραστηριότητες που είναι πολύ συχνά στις αναπτυσσόμενες χώρες. Από τα κάτι μέλη πρέπει να υιοθετηθούν δραστικά μέτρα για να υπάρξει ένα πρόγραμμα συνεργασίας με τρίτες χώρες, έτσι ώστε να διοργανωθεί σωστά η διασυνοριακή καταπολέμηση του ξεπλήματος. Πολλές φορές πρόκειται για περιβαλλοντικά ποινικά δικήματα, για φορολογικά, τα οποία ε, αναφέρονται στον κατάλογο που έχει προσαρτηθεί στο, στην έκθεση. Και παρουσιάζονται και στην πρόταση οδηγία της Επιτροπής. Κάτι που σημειώσαμε από τις μελέτες για τις αναπτυσσόμενες χώρες υπάρχει θέμα άγνοιας ε, γιατί δεν έχουν αρκετούς ανθρώπινους πόρους γιατί δεν μπορούν να έχουν την κατάλληλη ανακριτική μέθοδο αυτό είναι πολύ σημαντικό που να ενισχύσουμε εκεί τη συνεργασία μας Ιδίω για όσου από την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν μέσα και πείρα στην αντιμετώπιση αυτών των αδικημάτων. Η αντιμετώπιση λοιπόν αυτών των αδικημάτων παίρνει άλλη σημασία. Οι τροπολογίε τώρα 9 και 10. για το αδίκημα του ξεπλήματος. και την ε, ε, απόκτηση αγαθών. Αυτό δεν αφορά τόσο πολύ την Επιτροπή μας, αλλά περισσότερο τα, την πηγή του αδικήματος, δηλαδή τον τόπο που αυτό λαμβάνει η χώρα. Εάν δεν υπάρχουν όμως εργαλεία συνεργασία θα είναι αδύνατο αυτό για τους Ευρωπαίους δικαστές. Η τροπολογία 10 αφορά περισσότερο την εργασία τη επιτροπή ανάπτυξη. Εδώ δεν είμαι εγώ καθήλυνα αρμόδιο τη τη έκθεση. Προσπαθώ όμω να συντονιστώ με τον ε, αρμόδιο και για τη δουλειά αυτής της Επιτροπής και είμαι στη διάθεσή σας για να ακούσω οποιοδήποτε είδους προτάσεις θα μπορούσαν να βελτιώσουν το κείμενο που θα υποβάλουμε στα πλαίσια αυτής της έκθεσης. Ευχαριστούμε, Γκνάτσιο. Είναι πολύ σημαντικό γιατί θα πρέπει να κάνουμε κάτι, να πετύχουμε κάποια αποτελέσματα, αλλιώς δεν θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την ομοποίηση των παράνομων εισόδων. Ο Μπόγκταν είναι ο επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον Ιγνάτσιο, γιατί έκανε πραγματικά πολύ καλή δουλειά. Και πρέπει να πω ότι στην προετοιμασία της γνωμοδότησης για την οδηγία για την παρανομοποίηση του παράνομου χρήματος τα πήγε εξαιρετικά. Το σχέδιο αυτό είναι πολύ σημαντικό και για τη δική μας επιτροπή, ε, την Επιτροπή ΔΕΒΕ και κυρίως για τα θέματα συνεργασίας με τρίτες χώρες. Πιστεύω πως όλοι γνωρίζουμε τι γίνεται με τις τρομοκρατικές επιθέσεις εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και για να καταπολεμήσουμε τρομοκρατία θα πρέπει να στερήσουμε από τις τρομοκρατικές ομάδες ε, τις πηγές χρηματοδότησης που έχουν. Επίσης θα πρέπει να είμαστε σε θέση να εντοπίσουμε την χρήση από τις οργανώσεις αυτές παράνομων ε, μεθόδων πλουτισμού και αυτό αποτελεί ένα κομβικό στοιχείο τη στιγμή της καταπολέμησης της τρομοκρατίας όπως επίσης και του οργανωμένου εγκλήματος. Θεωρώ πως χρειάζεται κατεξουσιοδότηση πράξη η οποία θα προσπαθήσει να εντοπίζει τις τρίτες χώρες οι οποίες θεωρούνται υψηλού κινδύνου και νομίζω ότι εδώ δεν πρόκειται να καταγγέλουμε και να κατηγορούμε. Όχι, είναι επειδή ακριβώς θέλουμε να εντοπίσουμε ποιες είναι οι δικαιοδοσίε με τις οποίες είμαστε έτοιμοι και μπορούμε να συνεργαστούμε. Και αν υπάρχει βούληση συνεργασίας και από την άλλη πλευρά, τότε θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε και τις δυνατότητες που μας δίνει η αναπτυξιακή βοήθεια. Και ο κατάλογος αυτός δεν θα έχει να κάνει μόνο με τον περιορισμό των οικονομικών ε, σχέσεων με κάποια χώρα, αλλά το αντίθετο ακριβώς. Και χάρη στον κατάλογο αυτό πιστεύω πως θα μπορούσαμε με πιο αποτελεσματικό τρόπο να ελέγξουμε την κατάσταση. Η Ethereum οι επιχειρηματικοί εταίροι που συνεργάζονται με τη χώρα αυτή θα έχουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στα όσα συμβαίνουν στη χώρα και νομίζω πως αυτά ευθυγραμμίζονται και με τους στόχους που έχουμε θέσει, δηλαδή τη συμμόρφαση με μια σύσταση ε, της ε, ειδικής ομάδας εργασίας για την νομοποίηση παράνομων εσόδων ε, και τα σχετικά από την Επιτροπή ε, για τα θέματα αυτά. Άλλοι συνάδελφοι θέλουν να πάρουν το λόγο για το σημείο αυτό. Όχι. Τότε θα δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε τον κύριο Μπέντο Σίλβα από τη Γενική Διεύθυνση Home και τον κύριο Αλσίνα που επίσης είναι από τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων DG Home. Είμαι αναπληρωτής προϊστάμενος μονάδας για την αντιδημοκρατία στην ε, Γενική ε, Διεύθυνση Ιστορικών Υποθέσεων και χαίρομαι που έχω την ευκαιρία αυτή να πω δύο λόγια. Λέγομαι Μπέντου Σίλβα. Πιστεύουμε πως είναι πολύ σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση να κλείσει τη χρηματοδότηση μέσω ξεπλήματος. Έχουμε σχέδιο δράσης. Είναι από τις ε, κύριες προτεραιότητες στην Ένωση για την Ασφάλεια και για τα διαδικαστικά να σας πω πως θεωρούμε πως το τρέχον καθεστώς για ε, το ξέπλυμα δεν είναι επαρκώς αποτελεσματικό, δεν είναι αρκετά ενιαίοι οι ορισμοί στα κράτη-μέλη και επίσης δεν θα περιγράψω εδώ το περιεχόμενο της πρότασης, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Και λόγω της προσπάθειας που έχει κάνει ο συνάδελφός σας. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορώ εγώ να εκφράσω την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ενδεχομένως κάποιες τροπολογίες που θα λάβουμε, αλλά μπορώ να στείλω ένα μήνυμα και να σας πω πως παρακολουθούμε τα πράγματα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Βλέπουμε να είναι πολύ υψηλή ποιότητα οι εργασίε που κάνετε στι διάφορε επιτροπέ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αυτό χάρη στην πολύ συνεκτική προσπάθεια του εισηγητή, την πολύ καλά ε, τεκμηριωμένη μελέτη και νομίζω ότι έτσι αντιμετωπίζετε θέματα αυτά εδώ στο Κοινοβούλιο και όσον αφορά την έκθεση αυτή αλλά και τις επικείμενες ε, προτάσεις μας. Ένα τελευταίο. Για τα όσα είπε ο Πολωνός Ευρωβουλευτής. Αναφέρθηκε στον ε, ε, στην τρομοκρατία και τόσο θα κάνει και το Συμβούλιο Ασφαλείας ε, και η Ομάδα Εργασίας. Ναι, πολύ σημαντικά. Γιατί η προέλευση των ε, χρημάτων έχει να κάνει με την επικίνδυνότητα, αλλά ο κίνδυνος δεν είναι μόνο η καταχρήση, η φοροδιαφυγή και η φοροπαφυγή, αυτά που συνήθως ε, συνδέει κανείς με την νομιμοποίηση παράνομων εισόδων, πολλές φορές συνδέονται και με τη χρηματοδότηση των τρομοκρατικών επιθέσεων και οργανώσεων και γι' αυτό με ιδιαίτερη ικανοποίηση διαπιστώνουμε ότι η Επιτροπή σας εξετάζει και αυτή τη διάσταση με ένα πιο ολιστικό τρόπο δηλαδή για τα όσα συμβαίνουν στον χώρο της ασφάλειας. Όπως ακριβώς κάνουμε και εμείς. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Θέλει ο συνάδελφος να πει κάτι, όχι. Μία ερώτηση δική μου, γιατί δεν γνωρίζω τη σχετική νομοθεσία. Είναι η ΛΥΜΠΕ αρμόδια για το πώς θα λειτουργήσουν όλα αυτά επί τόπου. Εμείς καταλαβαίνουμε πως αυτή τη στιγμή πολλά παράνομα έσοδα χρησιμοποιούνται για την απόκτηση ακινήτων στις πρωτεύουσές μας. Δηλαδή μεγάλες επενδύσεις, κονδύλια που έρχονται, που αγοράζουν ακίνητα όπως επίσης και το πρόβλημα χωρών που ουσιαστικά δίνουν διαβατήρια σε ανθρώπους που επενδύουν στη χώρα τους. Και εκεί γνωρίζουμε πως δεν υπάρχουν αρκετοί έλεγχοι για το από πού προέρχονται τα κονδύλια αυτά τα οποία επενδύονται. Ξέρω πως έχουν σφίξει κάπως οι διατάξεις, γιατί εγώ πληρώνουμε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συνέχεια η τράπεζά μου μου ζητάει πληροφορίες γιατί να μου στέλνουν αυτές τις μεταφορές, τα εμβάσματα από το εξωτερικό. Όμως θα πρέπει να ανοίξουμε τα μάτια και να δούμε τι γίνεται και στις χώρες μας. Πολλά χρήματα κυκλοφορούν μέσα στο σύστημα και θα μπορούσαμε να κάνουμε περισσότερε ερωτήσει για το πού προέρχονται και ποιοι είναι αυτοί. Και νομίζω ότι πολύ σωστά λέω πως η χρηματοδότηση κατασχέθηκε στο προ... παρελθόν από προηγούμενους, από παλαιότερους ηγέτες ακόμα είναι κολλημένοι σε τραπεζικούς λογαριασμούς και δεν έχουν επαναπατριστεί. Οπότε πολλές φορές εμείς εντοπίζουμε την απάτη, το ξέπλυμα κτλ. Αλλά το να επιστρέψουμε τα χρήματα αυτά στους πραγματικούς ιδιοκτήτες κατόχους δεν γίνεται. Θα το αντιμετωπίσετε, υπάρχει αντίδραση από τα κράτη-μέλη όταν το προσπαθείτε. Ε, κυρία Κάτολα, το Αν έχω την ευκαιρία, θα ήθελα και εγώ να κάνω μια ερώτηση προ ε, τον εισηγητή και την Επιτροπή. Τι είναι, ποια είναι τα βασικά εμπόδια τώρα σε ό,τι αφορά τον εντοπισμό των δικαιούχων, των ιδιοκτητών. Αυτό θα είναι το βασικό ζήτημα και νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε πού βρισκόμαστε στο σημείο αυτό η Πρόεδρος. Αυτό το θέμα της ιδιοκτησίας την οποία έχουν τα καταπιστεύματα και όποιος άλλος και κανείς δεν ξέρει τελικά ποιος είναι ιδιοκτήτης αποτελεί ένα ζήτημα ομολογουμένως. Συγκεκριμένες ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μετά θα δώσουμε το λόγο και πάλι στον εισηγητή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Άντρε Στέφανο από την Γενική Διεύθυνση Home Task για την ε, Ένωση της Ασφάλειας, αλλά εκπροσωπώ και τη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης Justice, η οποία επίση έχει αρμοδιότητα τα αιτήματά σας είναι πολύ επίκαιρα. Φυσικά αυτό το εργαλείο απευθύνεται και προσπαθεί να επιλύσει ένα τμήμα του προβλήματος, το εγκληματικό κομμάτι αν θέλετε, όταν αποδεικνύεται ότι υπάρχει εγκληματική προέλευση των χρημάτων και ότι η διεκτησία αποτελεί τελικά το τελικό αποτέλεσμα χρημάτων που ξεπλένονται και εισαγάγονται στο οικονομικό σύστημα, ναι, θα υπάρχουν με το εργαλείο αυτό λύσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Γιατί τι συμβαίνει τώρα. Σε διάφορα κράτη-μέλη υπάρχουν διάφορα κίνητρα σε ό,τι αφορά τη φυλάκιση, σε ό,τι αφορά αποδεκτικά στοιχεία. Όταν θα, απο... θα εγκριθεί αυτό το μέσο, θα είναι πολύ πιο απλό για τους εισαγγελείς λόγω εναρμόνισης. Για παράδειγμα, στην Ισπανία να ζητήσει τη βοήθεια των ε, συναδέλφων του από τη Βουλγαρία, από την Ιταλία, για να συλλέξει αποδεκτικά στοιχεία. Αυτό είναι ένα από τα βασικά στοιχεία τα οποία προσπαθούμε να επιλύσουμε εδώ. Αλθεύει βέβαια ότι βασιζόμαστε στις ε, συνθήκες που έχει θέσει το Συμβούλιο της Ευρώπης. Τα κράτη-μέλη λογικά, μιας και ήδη έχουν προσπογράψει στη συνθήκη του Συμβουλίου της Ευρώπης, ε, θα θεωρούσαμε ότι είναι ήδη σε μια φάση εναρμόνιση, αλλά δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Χρειάζεται λοιπόν εναρμόνιση. Αλλά αυτό ασφαλώς αποτελεί και μόνο ένα κομμάτι του παζλ. Υπάρχει και το θέμα του δικαιούχου και του ιδιοκτήτη. Αυτό πάει χέρι-χέρι με μια άλλη διάσταση, την οδηγία κατά του ξεπλήματος χρήματος. Εγκρίθηκε το 2015, το 2017 τον Ιούνιο. Υποτίθεται ότι θα είχε μεταφερθεί στην Εθνική Νομοθεσία μέχρι τον Ιούνιο 2017. Δεν έχει γίνει η μεταφορά σε όλα τα κράτη-μέλη στις εθνικές νομοθεσίες. Τώρα προσπαθούμε να τροποποιήσουμε και την οδηγία. Είμαστε στον 5ο, 6ο, 7ο τριμερή διάλογο για την τροποποίηση της ε, οδηγίας. Τα θέματα τα οποία προσπαθούμε να τροποποιήσουμε στην οδηγία έχουν να κάνουν με τα είδη ιδιοκτησίας, τα οποία εξετάζουμε, οντότητες που θα πρέπει να επιδείξουν δέουσα επιμέλεια σε ό,τι αφορά τους πελάτες και καλύτεροι όροι για τον καθορισμό του ιδιοκτήτη και του δικαιούχου. Το εργαλείο αυτό λοιπόν στα πλαίσια της τέταρτης οδηγίας κατά της, ε, του ξεπλήματος χρήματος θα βοηθήσει ακριβώς το σημείο αυτό. Σε ό,τι αφορά και τις τράπεζες, τα χρηματοδοτικά ιδρύματα και άλλες τέτοιες ε, οντότητες στα πλαίσια της δέουσας επιμελίας. Ευχαριστώ πολύ η Επιτροπή Οίκων, φαντάζομαι την αρμόδια για την ε, καταπολέμηση του ξεπλήματος ε, χρήματος. Η Οίκων και η Λίμπα από κοινού ε, κάνουν τις διαπραγματεύσεις. Ιγνάσιο, μήπως έχεις να μας πει δύο λόγια για την πολιτική κατάσταση. Ναι. Για την οδηγία κατά του ξεπλήματος, εδώ συμμετέχει και έκον Πολύς χρόνος χάθηκε διότι η ΕΚΟΝ ήθελε να αναλάβει την έκθεση ε, και πριν η διάσκεψη των Προέδρων την αναθέσει και στην ΕΝΒΗ. Ε, και έτσι πρέπει να πιεστούμε λίγο χρονικά. Σωστά μα τα είπε ο εκπρόσωπο τη Επιτροπή εδώ. Ο στόχο είναι να υπάρξει εναρμόνιση των ποινικών συστημάτων. Αυτό σημαίνει ότι σήμερα στα διάφορα κατημέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν διαφορετικοί ε, τρόποι να καταλαβαίνει κανεί το ίδιο πράγμα, την ίδια υπόθεση. Οπότε, ανάλογα με την νομική κουλτούρα, την νομική. Ε, παράδοση στο κάθε κράτο μέλο, αντιμετωπίζεται διαφορετικά το ξέπλυμα του βρώμικου χρήματο και κάποια πράγματα δεν αναγνωρίζονται σε άλλα κράτη-μέλη. Θα μπορούσα να δώσω πολλά παραδείγματα. Λίγο χάρη στην Ιταλία υπάρχουν εργαλεία για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματο, τα οποία έχουν δημιουργηθεί για να καταπολεμηθεί η πραγματική καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματο τη μαφία στην Ιταλία άρχισε να δίνει καρπού τη στιγμή που άρχισαν να χτυπάμε απευθεία στα κεφάλαιά του. Ε, εργαλεία για το πάγωμα ή τη δίμευση των ε, κεφαλαιοσιακών, των κεφαλαιακών περιουσιών όσων είχαν εγκληματική δράση και το ξέπλυμα στην οικονομία των ε, ε, παράνομων αυτών εσόδων ήταν το μόνο αποτελεσματικό μέτρο. Σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες αυτό το εργαλείο σιάζει τελείως από το σύστημά τους. Υπάρχουν λοιπόν εκατομμύρια ευρώ τα οποία επενδύονται το είπατε, Πρόεδρε, σε όσα, με όσα συνέβησαν στο Λονδίνο, λόγου χάρη, ή σε άλλες χρηματαγορές για τα νομικά συστήματα πολλών ευρωπαϊκών χωρών δεν τίθεται καν το ερώτημα της προέλευσης αυτών των κεφαλαίων. Η οδηγία λοιπόν αυτή αναλαμβάνει διαφορετική σημασία διότι επιδιώκει να δημιουργηθεί ένα εσωτερικό νομικό σύστημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που να έχει κοινά σημεία αναφορά Να δίνει στου δικαστέ που είναι στην Ισπανία, την Ιταλία, τη Φιλανδία, τη Γερμανία, την Πολωνία περίπου το ίδιο εργαλείο αναφορά. Δηλαδή πέραν της συνεργασίας που ήδη υπάρχει και μιλάμε για τα εργαλεία δικαστικής συνεργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, θέλουμε μια οδηγία που να επιτρέπει το ίδιο πλαίσιο αναφοράς. Να καταφέρει να πλήξει τα ίδια τα κεφάλαια. Εμείς θα, θα προσπαθήσουμε να χρησιμοποιήσουμε ως σημείο αναφοράς όσα έχουν γίνει στην πράξη και έχουν χρησιμοποιηθεί ως εργαλεία και έχουν δώσει τα καλύτερα αποτελέσματα. Θέλουμε να χτυπήσουμε απευθεία τα παράνομα κεφάλαια. Αυτό ήταν το εργαλείο που εμεί είδαμε να λειτουργεί καλύτερα και αυτό το στόχο έχουμε χαθέσει στην οδηγία. Από την πλευρά των αναπτυσσόμενων χωρών, αυτό είναι ένα άλλο σκέλος, τα κεφάλαια που έρχονται απ' έξω, τα οποία είναι πιο δύσκολο να τα ανοιχνεύσουμε, εάν δεν υπάρξει και ένα σύστημα εσωτερική συνεργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Πρέπει εκεί να χρησιμοποιήσουμε παραμέτρους που στην περίπτωση των ανακριτών μας θα ε, κάνουν να ενεργοποιούνται τα ραντάρ. Δηλαδή μόλις ήταν κεφάλαια στο δικό μας, δικό μας σύστημα, στη δική μας αγορά, ε, θα έχουμε και θέματα τριβές ανταγωνιστικότητας ε, με ε, στην εσωτερική αγορά. Δηλαδή κάποιο που θέλει να ξεκινήσει μια οικονομική δραστηριότητα και θα ανταγωνιστεί κάποιον που παίρνει κεφάλαια από ξέπλυμα βρώμικου χρήματο εκτό λόγω εμπορίου ή διακίνηση όπλων λόγω χάρη περιβλητικών εγκλημάτων. Ε, είναι θέμα ανταγωνιστικότητα. Δεν μπορούμε λοιπόν να τα κάνουμε όλα αυτά ε, ε προστατεύοντα ε, μόνο όσου δρούν παράνομα και αφήνοντα απροστάτευτου αυτού που είναι νόμιμοι. Και για να γίνει αυτό πρέπει μια στιγμούλα να σκεφτούμε και την δική μας τη δικαστική κουλτούρα και να την ενισχύσουμε. Δεν μπορούμε μόνο να είμαστε ε, μανιώδεις των τεκμηρίων και να λέμε μόνο αν υπάρχουν σίγουρες αποδείξεις θα κάνουμε κάτι. Όχι. Ε, ε, να αντιστρέψουμε το βάρος της ευθύνης. Εσύ να μου αποδείξεις ότι το κεφάλαιο που διαθέτεις είναι νόμιμο, ε, προέρχονται από νόμιμες πηγές. Στην Ιταλία αυτό έχουμε πετύχει και αυτό δημιουργεί μια νομική κατάσταση διαφορετική. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε. Okay, so it's a very important piece of legislation, particularly in hand with the anti-money laundering directive revision, because that, only that one can tackle money. Εδώ πρέπει να το δούμε με προσοχή αυτό, διότι όντω μιλάμε για παράνομο χρήμα που έρχεται απ' έξω. Ε, και ήδη πρέπει εσωτερικώ ε, οι νόμοι δικοί μα να είναι συντονισμένοι. Ίσως να μην είναι θέμα αυτής της νομοθεσίας ε, το τι γίνεται εκτός, αλλά σίγουρα άπτεται. Ε, σας ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ που ήρθατε, ευχαριστώ για τις εξηγήσεις σας. Η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι στις 7 Σεπτεμβρίου το μεσημέρι. Και επειδή ε, βγάλαμε ένα σημείο από διάταξη, έχουμε 20 λεπτά παραπάνω διάλειμμα. Ψηφίζουμε στις 3. Ακριβώς. Και έχουμε μακροσκελή κατάλογο νομίζω, ε. Με πολλές συμβαστικές ε, ελπίζω. Θα σας δω και πάλι στις 3. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τους διερμηνείς.